Καλησπέρα συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την ε, Διακοινοβουλευτική Επιτροπή ε, η οποία γίνεται λόγω της ε, ετήσιας ημέρας για την βία κατά των γυναικών και θα μιλήσουμε για τη σύμβαση της, Κωνσταντινούπολη, της Κωνσταντινούπολης η οποία μιλά για τη βία κατά των γυναικών και συνεχίζω στη γλώσσα μου. Ε, χαίρομαι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και έχουμε αυτή τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε εκπροσώπους από 15 κράτη-μέλη και από την Νορβηγία. Επίσης έχουμε και από το Συμβουλίο της Ευρώπης, από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκπροσώπους. Θα ακούσω με μεγάλη χαρά την συνεισφορά όλων. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και όλα τα όργανα ε, και όλοι μαζί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βίας κατά των γυναικών μέσα από την προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Προσπαθούμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την πάταξη της βίας κατά των γυναικών με αυτή τη σύμβαση. Υπάρχει μια έκθεση και πολλές ε, δημόσιες ερωτήσεις που, έχουμε απευθύνει στην Κομισιόν το Σεπτέμβριο. Επίσης υπάρχει μια έκθεση για τη διαδικασία προσχώρησης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Επίση έχουμε και την, ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια και έχουμε ακούσει τη δική τους φωνή. Μια παρατήρηση για σήμερα. Να πω ότι η διερμηνία είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τα Ιρλανδικά και τα Δανέζικα. Επίσης υπάρχει μετάδοση της συνεδρίασης μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητές στον κατάλογο των ομιλητών και θα ήθελα να είστε σύντομοι. Θα σας ζητήσω λοιπόν ε, να το κάνετε αυτό, όπως επίσης και να συμπληρώσετε ε, ακριβώς ε, το έγγραφο που έχετε στο φάκελο που σας έχουμε δώσει, το φύλλο, το οποίο θα πρέπει να δώσετε μετά στην γραμματεία. Το θέμα μας λοιπόν είναι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη-μέλη, προσχώρηση και follow-up. Η κυρία Βυργίνια Λάγκμπαρκ, διευθύντρια από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα μας μιλήσει για τις μελέτες που έχει κάνει ε, το συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι για εμάς ε, είναι μια πραγματικά σημαντική ευκαιρία και στιγμή διότι έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, το 2013, όταν ήμασταν μόλις 2,5 ετών ως Ινστιτούτο, δημοσιεύσαμε την πρώτη πρόταση σχετικά με το τι μπορεί κανείς να μετρήσει όσον αφορά στη βία κατά των γενικών. Αν θυμάστε, ήταν τελείως κενό. Ε, πρώτον, δεν υπήρχαν δεδομένα για να συγκρίνουμε ε, ή επειδή η βία κατά των γυναικών ήταν και το αίτιο της ανισότητας των φύλων, επειδή υπάρχει η υπερίσχυση των αντρών εναντί των γυναικών, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και το αποτέλεσμα της ανισότητας των φύλων. Όταν φτιάξαμε το ίντεξ, είχαμε ήδη κάποια δεδομένα, είναι τα μόνα που έχουμε από την έρευνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέλαμε εκεί να διερευνήσουμε τι σημαίνει ενδοσυγική βία. Φέτος αναλύσαμε λίγο περισσότερο το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια σειρά μέτρων και μετρήσεων για να μετρήσει την πρόοδο σε σχέση με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και με τις ακραίες μορφές βίας που είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να μπορούμε να τις μετράμε. Τα προτείναμε, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε ακόμα καταφέρει αυτές τις μετρήσεις. Χρειαζόμαστε πολιτική δέσμευση, συμφωνία και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα χωρίς αυτά. Το του δείχνει ότι αν είχαμε κάνει μια τέτοια έρευνα ως τώρα, το επίπεδο αποκάλυψης πληροφοριών θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Η συνάδελφος Μπλαντίν θα σας πει σήμερα το πώς και το τι προτείνουμε να μετρήσουμε θεωρούμε ότι πραγματικά πρέπει να ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Ε, ευχαριστώ Βιργινία, για αυτή την ε, εισαγωγή. Νομίζω ότι πάμε καλά ως τώρα. Εγώ έτσι συνήθως ξεκινώ τη μέρα μου. Συνήθως ε, διαβάζω τις ειδήσει το να ξεκινάς ε, την ημέρα σου με τις ειδήσει όταν ασχολείσαι με αυτά τα θέματα που ασχολούμαι εγώ είναι ταυτόχρονα καλή και κακή ιδέα. Ε, διότι υπάρχουν ένα σωρό ε, για το πώς οι γυναίκες γίνονται θύματα, θύματα ξυλοδαρμού και βίας και στη συνέχεια δολοφονιών. το θέμα δεν είναι ε, το κατά πόσο οι άντρες ή οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μόνο, ε, η μέτρηση των ανισοτήτων είναι ένα πρώτο βήμα προς την περισσότερη ισότητα. Είναι ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε επαρκείς πολιτικές, να τις εφαρμόσουμε και να τις παρακολουθήσουμε. Αυτή λοιπόν η έννοια της μέτρησης των ανισοτήτων για να μπορέσουμε να πατάξουμε τη βία είναι ο λόγος που φτιάξαμε αυτόν τον ε, δείκτη της ισότητας των φύλων. Η βία ήταν εκεί από την αρχή, όμως δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε λόγω έλλειψης δεδομένων. Θα σας παρουσιάσω τώρα ένα πλαίσιο μέτρησης, μια πρόταση για τη μέτρηση της βίας και για να κατανοήσουμε το φαινόμενο, αλλά και για να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο της ισότητας των φύλων. Ε, έχουμε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο που βλέπετε εδώ, το βαθύ καφέ, είναι μια σειρά δεδομένων που αφορά στις πιο κοινέ μορφές βίας κατά των γυναικών. Αυτές που έχουν ποινικοποιηθεί, αλλά και αυτές για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα στις χώρες μας. Αυτά τα δεδομένα θα τα συγκεντρώσουμε και θα φτιάξουμε ένα σύνθετο μέτρο για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε μια περίπλοκη πραγματικότητα που έχει πολλές πτυχές και να την εντάξουμε σε ένα μέτρο για να ευαισθητοποιήσουμε και να παρακολουθήσουμε στο χρόνο και στο χώρο. Σε αυτό το στάδιο βέβαια αυτό δεν θα ήταν αρκετό, δεν θα μας δώσει μια συνολική εικόνα του φαινομένου. Γι' αυτό πάμε στο δεύτερο επίπεδο, τους επιπλέον δείκτες ε, που περιλαμβάνουν τις μορφές βίας που περιγράφονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πολύ σοβαρές μορφές, αλλά δεν μετρώνται επαρκώς. Ακροτηριασμός, ας πούμε, των ε, γυναικείων γεννητικών οργάνων. Δεν έχει ε, μετρηθεί αυτό με συγκριτικό τρόπο. Για κάποιες ε, μορφές ε, βίας ε, η ποινικοποίηση δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Και μετά έχουμε το τρίτο επίπεδο που είναι οι παράγοντες που έχουν να κάνουν με το ευρύτερο πλαίσιο για να κατανοήσουμε τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση της βίας και για να δούμε μέχρι πού φτάνει αυτή. Αυτά τα επίπεδα ορίζονται λόγω των υποχρεώσεων που έχουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη της Σύμβασης ε, τη Κωνσταντινούπολη. Για να παρακολουθήσουμε λοιπόν ε, τις τάσεις στην πάταξη της βίας. Άρα ποια είναι ε, η τάση, να έχουμε περισσότερη ποινικοποίηση της καταδίωξης του stalking δηλαδή και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Χρειαζόμαστε απαντήσεις και αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε. Και αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο θα βασιστεί σε διοικητικά δεδομένα κυρίως. Περνάμε τώρα ε, στα ιδιαίτερα στοιχεία του συνολικού αυτού μέτρου που ο στόχος του είναι να έχουμε ένα σκορ που θα μας δίνει σε ένα στιγμιότυπο το βαθμό της βίας που έχουμε σε κάθε χώρα. Και έτσι θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε και τις χώρες σύν χρόνο. Έχουμε λοιπόν ε, έναν ε, τριπλό στόχο. Καταρχάς, να μιλήσουμε για την επίπτωση της βίας, σωματική και σεξουαλική, αλλά και την γυναικοκτονία, που δεν περιλαμβάνεται και ούτε υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οπότε δεν μπορεί να υπολογιστεί προς το παρόν. Ο δεύτερος στόχος τώρα είναι να μετρήσουμε τη σοβαρότητα της βίας. Ποια είναι η επίπτωσή της στη ζωή των γυναικών. Και το τελευταίο είναι να μετρήσουμε την ετοιμότητα των γυναικών να συζητήσουν τη βία. Μιλάνε για την εμπειρία τους ή όχι. Ε, έχουν ε, κάποια πρόσβαση σε επαρκή προστασία από περαιτέρω βία. Σε αυτόν τον συνολικό δίκτυ, λοιπόν, σε αυτό το μέτρο, έχουμε συνδυάσει το σκορ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των δεδομένων ε, του Γραφείου των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπάρχει ένας δείκτης ισότητας ε, των φύλων. Μπορείτε να τον δείτε για να δείτε πώς είναι η χώρα σας, ε, που βρίσκεται. Αυτό λοιπόν το μέτρο ε, πηγαίνει από το 1 ως το 100. Αυτή είναι η κλίμακα. Όσο πιο υψηλό το σκορ, τόσο πιο μεγάλη ε, η επίπτωση ε, του φαινομένου της βίας. Τόσο πιο σοβαρή και κρυφή είναι η βία που συμβαίνει. Σε αυτό το πλαίσιο μέτρησης, λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο της βίας, το ενέκτασή της και να βρουν και μια μορφή προστασίας από αυτής και πάταξης αυτής. Για να καταλήξω θα σας πω ποια είναι τα συμπεράσματα που έβγαλε η ανάλυση μας. Καταρχάς, δεδομένα για τη γυναικοκτονία υπάρχουν μόνο στα μισά κράτη-μέλη και από το περιορισμένο αριθμό των δεδομένων και των χωρών μπορούμε να πούμε ότι κάθε μέρα μία γυναίκα χάνει τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της ή του πρώην συντρόφου της. Το 70% των θυμάτων είναι θύματα σωματικής και σεξουαλικής βίας και η βία οδηγεί σε επιπτώσεις στην υγεία. Καταλαβαίνετε πόσο τεράστιο είναι το κόστος οικονομικό και ανθρώπινο για τις κοινωνίες μας. Τέλος, ε, σχεδόν το ένα στα δύο θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκαλύψει την εμπειρία του σε κανέναν. Όχι στην αστυνομία, όχι σε γιατρό, όχι σε φίλους, όχι σε κανέναν. Δεν έχει αποκαλυφθεί αυτή η εμπειρία σε κανέναν και αυτές τις ημέρες αυτά προσπαθώ να έχω στο μυαλό μου γιατί ε, με όλες αυτές τις μαρτυρίες ε, και αυτό το ξέβρασμα της βίας ε, σκέφτομαι ότι ίσως ε, σιγά σιγά να υποχωρεί η σιωπή και να υπερισχύει η αποκάλυψη των πληροφοριών ε, διότι οι γυναίκες δεν ζούσαν στη ζωή τους χωρίς βία, απλώς ζούσαν με τη σιωπή. Και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αλλάξουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Βιργίνια Λάμπακ και την κυρία Μπλοντίν Μολάρ για τις παρουσιάσεις τους και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη Σιμώνα Λαντσόνη που είναι δεύτερη αντιπρόεδρος ε, της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της βίας ε, ε, κατά των γυναικών και κατά της ενδοοικογενειακής violence. Έχετε 7 λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Θα μιλήσω στα Ιταλικά γιατί είναι η πρώτη ευκαιρία που, την έχω, εφόσον, που έχω εφόσον υπάρχει διερμηνία και έχω σκοπό να την εκμεταλλευτώ. Όπως θα γνωρίζετε καλά, ε, μιλούμε για το όργανο παρακολούθησης ε, της Σύμβασης ε, της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αναφέρεται απευθείας στους θεσμικούς φορούς, φορείς με μιας χώρας σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να εναρμονιστούν οι διατάξεις της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας απέναντι στην σύμβαση στη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Το Μάρτιο υποβάλαμε το ερωτηματολόγιο το οποίο επεξεργάστηκε η αρμόδια επιτροπή το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα άρθρα της συμβάσεως. Το ερωτηματολόγιο αυτό διανεμήθηκε στην Αυστρία, τη Δανία και την Αλβανία. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την Τουρκία και το Μαροβούνιο και πολύ σύντομα από του χρόνου Σουηδία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Φιλανδία και άλλες χώρες. Κάτι που ε, επιτύχαμε ήταν ήδη να έχουμε 27 επικυρώσεις. Επομένως ε, φτάσαμε στο όριο των 25 επικυρώσεων. Και θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε πλέον την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα κρούσματα βίας από τα 10 στα 15 μέλη. τα μέλη του Γκρέβιο για να συμπεριλάμουν λοιπόν και άλλες χώρες Και ποια είναι τα πρώτα πράγματα τα οποία παρατηρήσαμε ή σημειώσαμε σε αυτές τις πρώτες παρακολούθησεις είναι παρακολουθήσεις, με συγχωρείτε, μόλις δημοσιεύσαμε τις σχετικές εκθέσεις για την Αυστρία και το Μονακό και σύντομα άλλες δύο θα έχουμε. Είναι δύσκολο λοιπόν να έχουμε μια τοποθέτηση με τη βάση τεσσάρων αναλύσεων, τεσσάρων χωρών. Όμως, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας επί διαφόρων ζητημάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο ερευματολόγιο, ένα από αυτά είναι και το θέμα των δεδομένων, στο οποίο αναφέρθηκε η Έγκεν, διοικητικά στοιχεία και δεδομένα, τα οποία θα μας επέτρεπαν να έχουμε μια πλήρη ερμηνεία για τα όσα συμβαίνουν σε κάποιο κράτος μέλος. Στον τομέα της δικαιοσύνης, ε, των αστυνομικών δυνάμεων, της υγείας, δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να συλλεχθούν και δύνατοι να συλλεχθούν ώστε να επικαιροποιείται αυτή η συλλογή, αυτά τα δεδομένα τα οποία θα μας επέτρεπε να διαμορφώσουμε πολιτικές, πώλησης λέει ο Μιλήτρια, διότι βασιζόμαστε αυτή τη στιγμή επί προβολών κυρίως, εκτιμήσεων. Όταν έχουμε λοιπόν δεδομένα και μάλιστα δεδομένα που θα είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους, αυτό θα μας επέτρεπε να διαμορφώσουμε, να κατευθύνουμε τις πολιτικές αντιμετώπισης των φαινομένων βίας κατά των γυναικών. Τώρα, το θέμα της ευθύνης που θα έχουν όλοι οι ενδιάμεσοι φορείς, ε, κρατικοί, δημόσιοι φορείς, το, θέμα της ε, δέουσας μέλειας αν θέλετε, ώστε να αποφεύγουμε κάποιες ερμηνείες που ενδεχομένως κάποιες φορές γίνονται με αυτοματοποιημένο και επιφανειακό τρόπο. και θα έλεγε κανείς μας χρειάζεται μια πολιτιστική επανάσταση, ριζική αλλαγή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε διατάξει σε όλα τα επίπεδα. Και χωρίς αυτήν την αλλαγή ε, αντίληψης, την πολιτιστική, πολιτισμική αλλαγή αντίληψης, θα είναι δύσκολο να βρούμε ακόμα και μια χώρα που θα έχει εναρμονίσει τις διατάξεις της έναντι τη συμβάσεω τη Κωνσταντινούπολη. Και προ την κατεύθυνση αυτή εργαζόμεθα. Βεβαίω εντό των διατάξεων πρέπει να εναρμονιστούν οι διατάξει αυτέ και έναντι του αστικού και ποινικού δικαίου, του αστικού και ποινικού κώδικα, ώστε να υπάρχει μια γραμμική συνέχεια. Υπάρχει όμως μια έντονη εστίαση, αυτό σίγουρα έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε επί της οικογενειακής βίας, αλλά και σε άλλα φαινόμενα και κρούσματα βίας που αναφέρονται ξεκάθαρα σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά που ακόμα δεν εξετάζονται στο ίδιο επίπεδο με την οικογενειακή βία. Και παρά την ιδιαίτερη αυτή υπογράμμιση, το θέμα των τέκνων καθίσταται σήμερα πρόβλημα η ίδια σύμβαση, το ίδιο, ο ίδιος φορέας του Γκρέβιο έχει κατηγορηθεί επανειλημμένος ότι, είναι, ότι στρέφεται κατά της οικογένειας, του θεσμού της οικογένειας. Λέω κατηγορηματικά ότι αυτό δεν ισχύει, δεν είναι αληθές. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία αντιθέτως πλήττουν το θεσμό και την παράδοση της οικογένειας και τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού. Το θέμα των τέκνων, όταν αυτά απομακρύνονται σε περιπτώσεις ε, κρουσμάτων βίας ή όταν αυτά μένουν απροστάτευτα, παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο παραμένει ανοιχτό πρόβλημα. το θέμα των επεμβάσεων, των βίαιων επεμβάσεων που υποχρεώνονται αρκετές γυναίκες σε διάφορα μέρη του κόσμου να υποβληθούν, το θέμα αδειών παραμονής και προσφύγων και συνδεδεμένων κρουσμάτων βίας, που είναι μία από τις βασικές θεματικές επί των οποίων υπάρχουν επιφυλάξεις από πλευρά κατών όπως και για το θέμα της αποζημίωσης των θυμάτων, το οποίο μας δίνει ένα συνολικότερο πλαίσιο των τάσεων ε, και κάπου εδώ νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει με τον χρόνο που έχω στη διαθέσή μου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Σιμώνα Λανσόνη και θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο στην Εύα Παστράνα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους ε, επαγγελματίες του νομικού τομέα του, HELP. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση αυτή. Εγώ είμαι υπεύθυνη του προγράμματος Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για την εκπαίδευση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για τους νομικούς επαγγελματίες, HELP, από εδώ και στο εξής. Και θα ήθελα σήμερα να σας πω ότι υπάρχει και ένα διαδικτυακό μάθημα ε, που αφορά την εκπαίδευση, στην προσπάθειά μας κατά πολέμηση της βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας. Ε, είναι ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο της προσπάθειας Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, για ποιο λόγο θέλουμε τώρα να το κάνουμε αυτό, γιατί αυτό λόγο θέλουμε να συνεργαστούμε. Ε, ο σκοπός του HELP είναι να βοηθήσει πράγματι ε, τους ε, δικαστές, τους νομικούς, τους εισαγγελείς να μπορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα εφαρμόζουν στην καθημερινή τους εργασία. Και η επιτυχία του HELP βασίζεται σε δύο συνιστώσεις. Πρώτον, είναι ένα δίκτυο ε, δικαστών, ε, συλλόγων ε, δικηγόρων, τεσσάρων χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως επίσης και άλλων εταίρων μας, όπως για παράδειγμα του Συμβουλίου Νομικών και Δικηγορικών Συλλόγων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η δεύτερη συνιστόσα είναι αυτά τα δωρεάν ηλεκτρονικά μαθήματα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα μας και τώρα ε, οι χρήστες της πλατφόρμας αυτής ε, έχουν ανέλθει σε πάνω από 20.000. Υπάρχει κατάρτιση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέσσερις φορές περισσότερους ε, χρήστες έχουμε σήμερα σε σχέση με πριν από τρία χρόνια. Τώρα, τι ζητούν οι άνθρωποι αυτοί και τι προσπαθούν να επιτύχουν μέσω αυτών των μαθημάτων. Ε, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρόσβαση ε, στους νομικούς επαγγελματίες και από εσάς και από διάφορους άλλους ε, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θέματος που θέλουμε να καλύψουμε σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όπως για παράδειγμα η μη διάκριση, προστασία των δικαιωμάτων, εργασιακά δικαιώματα, κακομεταχείριση, άσυλο, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, ε, εμπορία ανθρώπων, ε, άρχισε και έγινε και μια, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν από ένα μήνα και μια προσπάθεια που ξεκίνησε χθε για την επέτειο της Διεθνούς ημέρας κατά της βίας για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο θα το δημοσιευθεί, θα το ανακοινώσουμε δημοσίως κατά τις επόμενες ημέρες. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ των διαφόρων τμήματων ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, με το τμήμα ισότητας ε, ε, μεταξύ των φίλων ε, και του τμήματος του οποίου υπεύθυνη είμαι εγώ. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι μόνο παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, αλλά είναι και σοβαρή διάκριση κατά των γυναικών και μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως μόλις σας είπα, σεξουαλική κακοποίηση, σωματική βία, οικονομική πίεση, επίμονη παρακολούθηση, ακροτηριασμός ε, γεννητικών οργάνων ή εξαναγκαστική γάμη Το πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι να καταλάβουμε αυτό το είδος της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, ε, το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο με ιδιαίτερη εστίαση στην ε, σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης, στην οποία προσχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο στοιχείο, πώς μπορούμε να υπερβούμε τα εμπόδια που υπάρχουν για το να μπορέσουν να φτάσουν οι γυναίκες αυτές τη δικαιοσύνη. Επίσης, να υπάρχει μία ε, ποινική δικαιοσύνη και πριν από την ε, δίκη και μετά τη δίκη να υπάρχει μια ε, δίκαιη ποινή μετά τη δίκαιη δίκη Επίσης, να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Εδώ βλέπετε κάποιες απεικονίσεις οθόνης των ε, μαθημάτων που γίνονται ηλεκτρονικά. Η Bridget O'Laughlin είναι η γυναίκα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη της. Είναι εκτελεστική γραμματέας του Μηχανισμού Παρακολούθησης ε, του, της σύμβασης ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη σύμβαση συγγνώμη του Κωνσταντινούπολης, Συμβουλίου της Ευρώπης, αυτά τα μαθήματα δεν αφορούν μόνο τη μετάδοση γνώσης όσον αφορά το νομικό, ε, τη νομική γνώση. Θέλουμε να αλλάξουμε τις νοοτροπίες. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε και δεξιότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ε, έχουμε συμπεριλάβει πραγματικές ιστορίες, νομολογία, ε, υποθέσεις ορόσημα που έχουν διαμορφώσει την ευρωπαϊκή νομολογία ε, και από το Στρασβούργο αλλά και από το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Το διεθνές πλαίσιο υπάρχει, εστιάζει και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και, για το, και τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ε, όπως και άλλα μαθήματα του ε, HELP, του ε, προγράμματός μας. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, μπορείτε να δείτε εδώ για παράδειγμα τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μας λέει πόσο σημαντικό, ε, πόσο ε, καταστροφικά είναι τα ε, στερεότυπα γύρω από τα φύλλα και πόσο καταστροφική είναι αυτή η βία κατά των γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία και βίντεο διαφόρων εμπειρογνωμόνων όπως για παράδειγμα Γερμανού εισαγγελέα, Ιταλού δικαστή, Βούλγαρου δικαστή, ε, σε ένα, στο δικαστήριο του Στρασβούργου που ε, αγορεύει για ένα τέτοιο θέμα. Βλέπουμε λοιπόν ε, πώς ακριβώς έχει δομή των μαθημάτων. Σας εξήγησα τι στοιχεία περιλαμβάνει, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους χρήστες να καταλάβουν την ενδοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών. Και εδώ βλέπετε το δυναμικό της κάλυψής μας, μπορούμε να καλύψουμε 47 χώρες στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, όπου ε, ζουν 830.000 ε, άνθρωποι. Υπάρχει μία περιφερειακή προσέγγιση μερικές φορές όπως τα Δυτικά Βαλκάνια για παράδειγμα, στη Ρωσία, στην Τουρκία. Επίσης εστιάζουμε κάποια από τα μαθήματά μας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ολοκληρώνω την παρουσίασή μου επανεπισημένοντας ότι το HELP λειτουργεί, ε, υπάρχει όλο και περισσότερη ζήτηση για τα μαθήματα που προσφέρει και θα ήθελα να σας ζητήσω υποστήριξη προκειμένου να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα στα κοινοβούλια σας, ε, στα σχολεία, στους δικηγορικούς συλλόγους. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε επίσης ε, να μας βοηθήσετε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει περισσότερα χρήματα για την την ε, εκπαίδευση ως προς τα θέματα αυτά ε, καταπολέμησης της ε, βίας κατά των γυναικών, ενδοοικογενειακής βίας, και πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν μπορεί κανένας να το καταφέρει αυτό μόνος του. Υπάρχουν ε, αυξανόμενες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η αύξηση της ξενοφοβίας, ε, κοινωνική αδικία, ριζοσπαστικοποίηση, πολλά άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Να πω λοιπόν συμπερασματικά ότι πρέπει να πούμε ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου είναι λιγότερο από το 0,4% ε, και δεν το γνωρίζουν οι περί του συνολικού προϋπολογισμού. Δηλαδή από το συνολικό προϋπολογισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης μόνο το 0,4% πηγαίνει σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο και πιστεύω ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά και να επιφέρουμε πραγματικά ε, σοβαρά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση βίας κατά των γυναικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννα Πετρόφσκα τώρα, πρόεδρος ε, τη της, ε, ε, του Ιδρύματος Φεμινοτέκα για την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ ε, που μου δώσατε το λόγο. Θα ξεκινήσω ευθύ αμέσως γιατί δεν έχω χρόνο και έχω μια μεγάλη παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη για το γεγονός ότι η παρουσίαση είναι στα πολωνικά, όμως ζούμε δύσκολες στιγμές στην Πολωνία να εξηγήσω τα πράγματα που ήθελα να σας αναφέρω σήμερα το απόγευμα. Καταρχάς, σύντομα να μιλήσω για την κύρωση της σύμβασης ε, της ε, Κωνσταντινούπολης στην Πολωνία. Γιατί τα πράγματα δεν πήγαν τόσο μαλά. Οι οργανώσεις όπως και οι δικοί μου έπρεπε εξ αρχής να παλέψουν για την προώθηση της ε, εκπαίδευσης και της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης πόσο βοηθά στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και στην πάταξη της βίας. Ε. Θα σας πω τώρα και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κύρωσης και πώς προχωράει η εφαρμογή. Η Πολωνία υπέγραψε τη σύμβαση ε, το 2015. Ο πρόεδρος ε, κύριος Κομορόφσκι ε, την υπέγραψε και έκτοτε από τον Αύγουστο δηλαδή του 2016 είναι σε ισχύ. Αυτή εδώ είναι η φωτογραφία του Προέδρου ε, να υπογράφει, παρόλο που ο ίδιος είχε κάποιες επιφυλάξεις. Η πολέμα, οι πολέμοι της σύμβασης έλεγαν ότι η σύμβαση απειλεί την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τις ε, θρησκευτικές παραδόσεις της Πολωνίας. Φαίνεται ότι για αυτούς ήταν ε, αναγγελία πολέμου κατά της ε, πολωνικής κουλτούρας. Στην μίλησαν για μια ιδεολογική αναδιαμόρφωση του πληθυσμού. Έλεγαν ότι η ισότητα των φύλων είναι αιρετική ε, άποψη και δεν υφίσταται στην πράξη. Ο Πρωθυπουργό εκείνη την εποχή, ο Ντόναλτ Τούσκ, τράβηξε τη διαδικασία κύρωσης ε, της σύμβασης δεν υπήρχε πλειοψηφία. Ο Πρωθυπουργό Κόπετς είπε ότι θα υπερψήφιζαν τη σύμβαση, αλλά δεν μπορούσε να επιβάλλει την άποψή του στους ε, βουλευτές. Ο πρόεδρος Κομορόφσκι είπε ότι δεν τον ικανοποίησε πλήρως η γλώσσα της ε, σύμβασης, διότι δεν τέριαζε με τα κοινωνικά ήθη της Πολωνίας. Αυτό ε, ε, στην ουσία αναφερόταν στο λεξιλόγιο που έχει να κάνει με το ε, σεξ και με το φύλλο. Σύμφωνα με την νομοθεσία της Πολωνίας, η ειδική αναφορά στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών ε, δεν υφίσταται, δεν αναφέρεται η πολωνική νομοθεσία στις γυναίκες συγκεκριμένα και τα κορίτσια ως θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει μια κοινωνική διάσταση του φίλου και το γεγονός ότι η σύμβαση αναφέρεται σε στερεότυπα για το φύλλο ως αιτία κάποιες φορές της βίας κατά των γυναικών είναι κάτι που ε, στην ουσία δυσαρεστούσε τους ε, πολέμιους ε, των τη σύμβαση στην Πολωνία. Δυστυχώ η ομιλήτρια μιλάει πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσει να διερμηνευτεί σωστά. E, i konwencja Η σύμβαση ζητά τα αγόρια και οι άντρες ε, να μάθουν για τη βία κατά των γυναικών, να εκπαιδευτούν. Επίσης, επικεντρώνεται στα αίτια της βίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς και στα στερεότυπα για τις γυναίκες. απαιτεί ε, τα κράτη να αντιδράσουν και να δράσουν κατά της ε, ενδοοικογενειακής βίας. Χάρη στην κύρωση της σύμβασης από την Πολωνία, είμαστε τώρα σε θέση να δώσουμε και να έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη δίωξη του βιασμού. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο όφελος ε, αυτής της σύμβασης. Η Κακός καραγιά η οποία είναι βουλευτής, ε, ε, ήταν και η συνήγορος του πολίτη εκείνη την εποχή. Χάρη σε αυτήν λοιπόν και χάρη στη δική μου οργάνωση μπορούμε πλέον να έχουμε την προστασία των θυμάτων. Η καθηγήτρια Μαγκουζάτα Φουσάρα Επίσης έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην όλη διαδικασία της προστασίας των θυμάτων από την αστυνομία και στο δικαστήριο. Δεν έχει ακόμα βέβαια εφαρμοστεί πλήρως αυτό. Έχουμε όμως ε, μία ε, γραμμή ε, δωρεάν που μπορεί κανείς να καλέσει 24 ώρες το 24ωρο για να καταγγείλει τέτοια ζητήματα. Επίσης υπάρχει και ο ορισμός για την οικονομική βία, κάτι που δεν υφίσταται στην νομοθεσία της Πολωνίας. Η νομοθεσία μας επίσης και τα προγράμματα που έχουμε κατά της ενδοοικογενειακής βίας δεν αναφέρονται πουθενά σε βία λόγω του φύλου. Δηλαδή βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και αυτό δεν μας ικανοποιεί. Ζητήσαμε να διορθωθεί αυτό, να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Είπαμε ότι η νομοθεσία θα έπρεπε τουλάχιστον στο προήμιο να αναφέρει κάτι για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Μα ως τώρα δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξει δημόσια συζήτηση της σύμβασης στην Πολωνία, γιατί θα σας πω σύντομα τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μου. Przepraszam, ale Ζητώ συγγνώμη, αλλά φαίνεται ότι το μηχάνημα δεν με ακούει. Ωραία. Θα αφήσω αυτή την όμορφη φωτογραφία εδώ να βλέπετε και θα σας πω αργότερα τι ακριβώς ε, είναι. Να πω στο μεταξύ ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης χαιρετίστηκε από, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τουλάχιστον από αυτούς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που ήταν ευνοϊκά προσκύμενοι απέναντί μας. Και μάλιστα δώσαν κονδύλια για την εκπαίδευση, την πληροφόρηση, άλλαξαν τα κείμενά τους για να χρησιμοποιούν την φρασιολογία μας και σε πολλές περιπτώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση είχαμε επιτυχία στην Πολωνία. Ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή παλεύουμε, βλέπετε εδώ τον Κατσίνσκι, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ε, του νόμου και της δικαιοσύνης, Το Δεκέμβρη Αυτό το κόμμα έκανε κάποιες προσπάθειες ε, για να βγούμε από τη σύμβαση. Τελικά φάνηκε ότι τα επιχειρήματά του ήταν σαρθρά, μετά ε, ο πρόεδρος ε, είπε ότι δεν θα βγούμε από τη σύμβαση αλλά ούτε και θα την εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή που σας περιέγραψα. Είμαστε, απειλείται η σύμβαση και πολύ πιθανό η Πολωνία να βγει από τη σύμβαση. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τώρα. Θα θέλαμε να ακούσουμε από τις αντιπροσωπείες ε, και τα μέλη, αλλά έχουμε πλέον μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Λέει Πρόεδρος, θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω να είστε πολύ συγκρατημένη, πολύ σύντομη στι όχι περισσότερο από δύο λεπτά. Η κυρία Αριστίδου, παρακαλώ, από την Κύπρο. Παρακαλώ. please, Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδελφοί σας, η Κύπρος υπέγραψε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 2015 και την επικύρωσε τον Ιούλιο του 2017. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών διαδραμάτισε καταλητικό ρόλο στην κύρωση τη Σύμβαση, αναδεικνύοντα την επιτακτική ανάγκη επικύρωση τη Σύμβαση και εξυγχρονισμού τη νομοθεσία, προκειμένου να ανταποκρίνεται στι υποχρεώσει που απορρέουν από τη Σύμβαση. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ στι αξιοσημείωτε πρωτοβουλίε που ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνη στο πλαίσιο σταδιακή υιοθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση νομοσχέδιο που ποινικοποιεί την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση, όπω ορίζει το άρθρο 34 τη σύμβαση. Επίση, ετοίμασε νομοσχέδιο για ποινικοποίηση τη βία κατά των γυναικών, ώστε να ενσωματωθούν πλήρω οι πρόνοιε τη σύμβαση στο Κυπριακό Δίκαιο. Η προτινόμενη νομοθεσία εγκαθιδρύει ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και ενσωματώνει πρόνοιες για λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων τόσο προληπτικού όσο και κατασταλτικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, ο ρόλος της αστυνομίας αναβαθμίζεται ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη στην πρόληψη και στην άμεση ανταπόκρισή της στα περιστατικά βίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιχορήγηση σε αιτήσια βάση της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των θυμάτων βίας που λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια σε 24 ώρη βάση όπως προβλέπει και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης Καταλήγοντα, θα ήθελα να τονίσω ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου τη έμφυλη βία απαιτεί συνέργεια, συλλογικότητα και συντονισμό δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε κυβερνητικό και μη κυβερνητικό επίπεδο. Η κύρωση τη σύμβαση είναι η αρχή του δρόμου και όχι του τέλου. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ματέρα παρακαλώ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ήμουν σε άλλη επιτροπή γιατί έπρεπε να ψηφίσω. Ε, να συγχαρώ και εγώ για την προσχώρηση στην Σύμβαση Κωνσταντινούπολη, ε, η δουλειά του Γκρέβιο είναι απαραίτητη για να καταλάβουμε κατά πόσον οι διατάξει τη συμβάσεω αυτή θα υλοποιηθούν σωστά από τα κράτη-μέλη. Η επικύρωση των διεθνών συμφωνιών είναι συχνά μια δικασία αρκετά αργή συχνά υπογράφουν τα κράτη-μέλη για να ανταποκριθούν στι πιέσει των ε, κοινωνικών και ενδιαφερομένων φορέων, αλλά από εκεί και πέρα ε, μένουν ακόμα μακριά από την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. 23 είναι μέχρι σήμερα οι χώρες που έχουν επικυρώσει, μεταξύ των οποίων 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα καταλογοποιήσω για να μην μακρηγορώ. Και οι 14 αυτές χώρες έχουν απλώς υπογράψει τη σύμβαση, η οποία έχει νομικές επιπτώσεις άμεσης. Κάποιες χώρες πριν επικυρώσουν χρειάστηκε να προσαρμόσουν τον ποινικό τους κώδικα και άλλες διατάξεις κατά των κρουσμάτων βίας προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τον ορισμό και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στο πλαίσιο της βάσεως. Κάποιες άλλες καθυστερήσεις οφείλονται σε πολιτικούς και όχι τεχνικούς λόγους, όπως η αντιπαράθεση που έχει σχέση με την έννοια του φύλου, και τα στερεότυπα που συνδέονται με την ερμηνεία του. Οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή διαφωνία θα πρέπει να παραμεριστεί καθότι ο βασικός στόχος της συμβάσεως είναι να παρέμβει ε, με αποφασιστικότητα κατά των, κρουσμάτων βίας, ε, κατά των γυναικών, κατά των οικογενειακών κρουσμάτων βίας. Ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα διάφορα ψηφίσματα στα οποία προχωρήσαμε, ζητήσαμε από τα κάθε μελη να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατό τη σύμβαση και να προσχωρήσουν απολύτω στην συμφωνία χωρίς να τοποθετήσουν επιφυλάξει Και, και ολοκληρώνω. Νομίζω ότι η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη θα έπρεπε να συμπληρώσει και όχι να υποκαταστήσει τις προσχωρήσεις των μεμονωμένων κρατών μελών, η προσχώρηση δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, και να συμπληρώσει το πλαίσιο των θεσμικών υποχρεώσεων που διέπουν την προστασία των θυμάτων και επίσης θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια των εθνικών πολιτικών κατά των κρουσμάτων ε, οικογενειακής βίας και βίας κατά των γυναικών που τοποθετούνται στο εσωτερικό των, ε, της νομοθεσίας του κάθε κράτους μέλους. Και ήθελα να απευθύνω και ένα μικρό ερώτημα στην κυρία Λαντζόνη. αν με επιτρέπετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύετε ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να είναι ένα πραγματικό βήμα προς τα εμπρός προς την υλοποίηση της συμβάσεως και επίσης πώς διεξάγεται και πώς θα διεξαχθεί αυτή η παρακολούθηση, αυτή η επιτήρηση στην οποία αναφερθήκατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ματέρα, λέει η Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους ε, συμμετέχοντες στη συνεδρίασή μας ότι ήδη 17 κράτη-μέλη επικύρωσαν. Τελευταία ήταν Γερμανία, Εστονία και Κύπρος. Οι οποίες χώρες θα μπορούσαν να δώσουν το καλό παράδειγμα και στις υπόλοιπες θα έλεγα. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μαλντεκιένιε, μέλος του Λιθουανικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. υπάρχει άσκηση ε, αρκετής οργανωμένης πιέσεως και lobbying σχετικά με αυτήν τη σύμβαση, διότι υπάρχουν αρκετές αμφίσιμες διατάξεις. Η ερμηνεία της έννοιας gender θεωρείται επίθεση κατά των χριστιανικών αξιών. Και γι' αυτό εκφράζεται και μία αντίρρηση διαφωνία προς την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση όταν ε, υπησέρχεται το θέμα η εξέταση σε θέματα διαφοροποίησης φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Εγώ απερίφραστα υποστηρίζω τη σύμβαση και την επικύρωσή της, αλλά ε, με βάση τις αναλύσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή μια θετική ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, ως έχει το κείμενο. Θα πρέπει λοιπόν να διεξαχθεί μια συζήτηση προκειμένου να οδηγηθεί το θέμα στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας μας, ώστε να διευκρινίζεται αυτή η ερμηνεία που έχει δοθεί ότι πρόκειται για επίθεση κατά των βασικών αξιών του Λιθουανικού Συντάγματος. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπεσίρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλου του ε, συμμετέχοντε ε, στη σημερινή συζήτηση και ιδιαίτερα την κυρία Πιετρόφσκα, γιατί γνωρίζουμε την κατάσταση που αντιμετωπίζετε στην Πολωνία. Έχετε όλη τη στήριξή μας και έχετε την ε, υποστήριξή μας για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Θα σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε. Πρέπει να ποσοτικοποιήσουμε το πράγμα και να το αναλύουμε διαρκώς γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε σωστά. Και ποια είναι η εστίαση που έχουμε δώσει το θέμα μέχρι εδώ. Η εστίαση μας είναι επί των θυμάτων. Και αυτό είναι σωστό. Πρέπει να προστατεύουμε τα θύματα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η θυματοποίηση, για να το πω έτσι, που γίνεται μέσω της εστίασης αυτής, προχωρεί μαζί με την δημιουργία κάποιων ενοχικών αισθημάτων που ίσως να δημιουργούνται σχέση με το θέμα. Εμείς ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε επαρκώς το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προσπάθεια που έχει καταβάλει με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, γιατί είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό όργανο που έχουμε πλήρες για το θέμα αυτό και υπέρ της δίωξης αυτών που διαπράττουν αδικήματα στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, που προχωρούν δηλαδή σε... που ασκούν βία οικογενειακή κατά των γυναικών, ο οποίος μπορεί να είναι ένας βιαστής, ένας εκβιαστής, μπορεί να είναι μπορεί να λάβει πολλές μορφές αυτό το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να διαπράξει διάφορα ποινικά και άλλα αδικήματα στο πλαίσιο της σύμβασης και του ποινικού κώδικα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την δίωξη και την καταγγελία των φαινομένων αυτών, την δίωξη των υπευθύνων, για να αλλάξουμε λίγο τον προσανατολισμό μας. Ευχαριστώ κυρία Μπεσέρα. Η κυρία Πουτσουφλέσκα. Από το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ σήμερα. Εγώ έρχομαι από αυτήν την οπισθοδρομική, για να την πω έτσι, χώρα, την Πολωνία. Όπως είπε και η κυρία Πιοτρόφσκα, όντως η Πολωνία θέλει να αποσυρθεί από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η σύμβαση μας πάει πίσω στις 11 Μαΐου του 2011. Τότε ο Υπουργός ε, Εργασίας και Κοινωνικών Ζητημάτων ε, το Μάιο του 2011 πριν ε, την γένεση της συγκεκριμένης σύμβασης που μιλούσε υπέρ της υποστήριξης των θυμάτων. 35 κέντρα, ειδικά κέντρα αντιμετώπισης ε, των προβλημάτων αυτών και ε, βοήθειας των θυμάτων και θα υπάρξει άλλο ένα το 2019. Πρόκειται για εξειδικευμένα κέντρα ε, που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τα θύματα βίας. Κάθε τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχει ε, στον τομέα, ε, στην προσπάθεια αυτή. Και δεν είναι μόνο τα κορίτσια και οι γυναίκες ε, που είναι θύματα και άλλα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, όπως οι πιο ηλικιωμένοι, παιδιά, είναι συχνά θύματα βίας και Γι' αυτά ακριβώς τα θύματα ε, θέλει να φροντίσει το ε, Υπουργείο ε, Εργασίας, Υγείας, Κοινωνικών Ζητημάτων, Εσωτερικών, Εκπαίδευσης, Πολιτιστικής Κληρονομιάς. όλα αυτά τα υπουργεία έχουν ω μέλημα τους ανθρώπους αυτούς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν και καθήκον να ενημερώνουν και να μεταδίδουν ε, τις πληροφορίες σε σχέση με τους τρόπους πρόληψης της βίας. Θα θέλα λοιπόν να ζητήσω να μην λέγεται ότι οι Πολωνοί δεν θέλουν ε, να βοηθούν ε, τους ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό δεν είναι σωστό και δεν είναι και αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο χρόνος που αναλογούσε σε αυτή την πρώτη μας συζήτηση πλησιάζει στο τέλος του, οπότε δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώ δεν μπορώ να δώσω σε άλλους ομιλητές ε, το λόγο, ούτε να δώσω και στους προσκεκλημένους το λόγο να απαντήσουν θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε το λόγο στη δεύτερη συζήτηση, λέει ο πρόεδρος. Ή πρόεδρος, συγγνώμη. Εντάξει, να σας δώσω το λόγο, εφόσον δεν πήρατε το λόγο προηγουμένως. 1,5 λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει και εγώ να μεταβώ σε άλλη συνεδρίαση τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις συμμετέχουσες στη σημερινή συζήτηση και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια αφιέρωση σε μια νεαρή 18 χρονών που λέει ναι, εγώ πιστεύω. Una chica de 18 años. Στην Παμπλώνα πέρυσι, αν ακούσαμε καλά, ε, έγινε μια επίθεση πέντε ανδρών κατά της νεαρής αυτής. Είχαμε βίντεο που κυκλοφόρησαν WhatsApp και λοιπά Και τελικώς βλέποντας τις δηλώσεις που γινόντουσαν σχετικά με τον περιστατικό, κάποιοι τοποθετήθηκαν για να υποστηρίξουν την νεαρή αυτή και να πούνε ναι, εγώ σε πιστεύω. Η πρώτη έρευνα για τα κρούσματα αυτά βίας του 2015, στα πλαίσια της έρευνας αυτής, έγιναν, ερωτήθηκαν χιλιάδες άτομα στην Ευρώπη και αυτή η περίπτωση ανταποκρίνεται απολύτως ανάμεσα στις περιπτώσεις κρουσμάτων βίας. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε όλοι υπέρ της επικύρωσης από πλευρά των κρατών μελών της συμβάσεως, αλλά εδώ μας χρειάζεται πολιτική βούληση. Η επικύρωση κάθε αυτή δεν σημαίνει ότι τα κράτη θα επιδείξουν βούληση. Ούτε η μη επικύρωση απαγορεύει, παρεμποδίζει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν μέτρα υπέρ της ισότητας και της ισότιμης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Η υπέρ τη αντιμετώπιση των κρούσματων βία. Απλώ αυτή η σύμβαση σημαίνει ότι θα έχουμε κάνει ένα βήμα προ τα εμπρό. Συμβολικό βήμα. Αυτό που μα χρειάζεται και αυτό που εγώ ζητώ είναι πολιτική βούληση. Στην αυτονομία την βασική τα τελευταία δύο χρόνια εγκρίθηκαν δύο νομοσχέδια και παρόλα αυτά έχουμε τέτοια κρούσματα βίας στη χώρα μου, στην περιφέρειά μου. Πριν από 10 χρόνια η πρώτη ένωση που συναισθήθη στη χώρα των Βάσκων ε, έγινε δεκτή από το, Εθνικό, από το Κοινοβούλιο το Περιφερειακό και τότε όλοι μας είπαν και οι εκπρόσωποι της Βουλής και ο κόσμος ότι πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας. Βλέπουμε κάθε χρόνο κρούσματα φούνου παιδιών από γονείς οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από το σεξουαλικό τους προσανατολισμό μεταξύ άλλων. Δηλαδή οποιαδήποτε, οποιοδήποτε κρούσμα βίαιο πρέπει να οδηγεί σε μια αντίδραση. Σε μια αντίδραση οργανωμένη από την κοινωνία, από τους θεσμούς. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να παρατηρούμε να υποβιβάζουμε τα δικαιώματα του μισού πληθυσμού μας που είναι οι γυναίκες στον κόσμο αυτών και στις χώρες μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να επιτύχουμε επιτέλους την έκφραση της πολιτικής βούλησης των χωρών ώστε να λάβουν αυτά μέτρα κατά των κρουσμάτων βία και υπέρ τη ισότητα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει άμεσα να πάω σε άλλη συνεδρίαση και γι' αυτό ήθελα να μιλήσω τώρα. Ε, Ευχαριστώ την κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα και τώρα δίνω το λόγο στην τελευταία ομιλήτρια του πρώτου πάνελ, η κυρία Φατορίνη από την Ιταλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Εγώ, εμείς, ε, με συγχωρείτε, στην ε, Ιταλία ομοφόνο στο Κοινοβούλιο εγκρίναμε την επικύρωση αυτή, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική για δύο λόγους. Καταρχά είναι δεσμευτική νομικά, δεν είναι απλά μια ασαφής δήλωση ή διακήρυξη και δεύτερον διότι άπτεται του κεντρικού πυρήνα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ισότητας δηλαδή των φίλων. Και ήθελα για αυτό το λόγο να πω προς τις φίλες και τους φίλους από την Πολωνία και το λέω με το χέρι στην καρδιά λέει ο Μιλήτρια. Όλα αυτά δεν είναι απειλή κατά της οικογένειας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ο τρόπος για να ενισχύσουμε τους οικογενειακούς δεσμούς τους δεσμούς συντροφικότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτές οι σχέσεις εδράζονται επί της αμοιβαίας αξιοπρέπειας και σεβασμού. Είναι ακριβώς αυτές οι χριστιανικές καθολικές αξίες που οι συνάδελφοι από την Πολωνία φοβούνται ότι μπορεί να πλήττονται. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς αυτούς. Και το λέω. Γιατί εδώ δεν μιλούμε για κάποιες περιθωριακές απελπισμένες περιπτώσεις μιλούμε για κανονικότατες, για να το πω έτσι, οικογένειες, νοικοκυριά παντού στην Ευρώπη. Και εγώ θα μπορούσα να κατανοήσω σε μεγάλο βαθμό την ανησυχία σας, αλλά δεν πρέπει να φοβούμαστε την έννοια του φίλου, την έννοια του gender. Δεν σχετίζεται όμως αυτή καθε με την εμφάνιση, με την εμφάνιση των, των κρούσματων βίας. Διότι ε, ακριβώς εδώ βρίσκεται το κεντρικό ζήτημα της, του αμοιβαίου σεβασμού και αξιοπρέπειας στα πλαίσια ενός δεσμού, συντροφικού δεσμού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα έπρεπε να υγείστε της προσπάθειας αυτής και όχι το αντίθετο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για άλλη μία φορά όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησης και τώρα πάμε στο δεύτερο πάνελ το οποίο αφορά στην εφαρμογή της Σύμβασης της Ισταμπούλ σε εθνικό επίπεδο. Θα μιλήσουμε και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Δίνω λοιπόν ε, το λόγο του δώσω στους ευρωβουλευτές και τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων το λόγο. Δίνω το λόγο τους εκπροσώπους από την Ιταλία και την Ισπανία και από την κοινωνία των πολιτών. Yeah, Miss Francesca Puglisi. Hello. Hello. Hello. Thank you for coming. Nice to meet you. Miss Pilar Cancela Rodriguez. Κυρία Πιλάρ Cancela Rodriguez, είστε εδώ. Είναι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου, η, κυρία, η Ζακή Χάντ επίσης. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Πρώτη, η κυρία Φραντσέσκα Πουλίζη Πρόκειται για την πρόεδρο της, ε, Επιτρο... της Ανακριτικής Επιτροπής του, Ευρω... του Κοινοβουλίου της Ιταλίας ε, για την γυναικοκτονία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι είμαι η πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής της Ιταλικής Γερουσίας κατά των κρουσμάτων ε, βίας κατά των γυναικών και των δολοφονιών. Ήμασταν μεταξύ των πρώτων χωρών που επικυρώσαμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από τον Ιούνιο του 2013 και ήταν μία από τις πρώτες πράξεις της παρούσας ε, θητείας. Πράγματι στη δική μας ε, Βουλή έχουμε έναν σημαντικό αριθμό γυναικών και ακριβώς μετά την επικύραση της συμβάσεως ενεκρίθηκε το διάταγμα για τις γυναικοκτονίες με σημαντικά μέτρα δηλαδή συγκεκριμένε αποζημιώσεις για όσες καταγγέλουν, για όσε γυναίκε καταγγέλουν τέτοια φαινόμενα, μέτρα απομάκρυνση από την οικογενειακή αιστεία δραστών ή ενόχων, προστασία ανηλίκων. Ακόμα πιο σημαντικό για μια πραγματική αλλαγή στην κοινωνία μας, όπως ε, επικαλείται και η σύμβαση, στα σχολικά προγράμματα στο σημείο 16 του νόμου 107 προσθέσαμε το αίτημα σε όλα τα σχολεία τα οποία ενέχουν δράσεις για την εκπαίδευση των νεαρών και της νεαρές στοιχεία για την αποφυγή ε, κρουσμάτων βίας και για την ισότητα των φίλων αλλά και για την κατάρτιση των ίδιων των ε, δασκάλων το 2015 υπευλήθη το πρώτο έκτακτο εθνικό σχέδιο κατά της βίας μεταξύ των φύλων. Καταρχάς ώστε να υπάρχει ένας φορέας συντονισμού μεταξύ όλων των θεσμικών φορέων και κρατικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τα κρούσματα αυτά και ένα παρατηρητήριο που θα φέρνει σε επαφή και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τα κέντρα κατά της βίας μαζί με τις υπόλοιπες ε, κρατικές υπηρεσίες. Φέτος δημιουργήθηκε και αυτή η ερευνητική επιτροπή προκειμένου να παρακολουθήσει την υλοποίηση και την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων της Συμβάσεως Κωνσταντινούπολης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι 60 εκατομμύρια από το 2013 στο 2016 και η εφαρμογή των διατάξεων. Αυτά που προκύπτουν λοιπόν μετά από πάρα πολλές ακροαματικές διαδικασίες και παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει πολύ προχωρημένο νομοθετικό πλαίσιο, καθότι παρά το γεγονός μάλλον ότι κατέρχονται έντονα συνολικά ή τα κρούσματα δολοφονίας ή γυναικοκτονία δεν κατέρχεται. Μία γυναίκα δολοφονείται κάθε δύο ημέρες και κάποια μέτρα όπως η απομάκρυνση από την οικογενειακή αστεία χρησιμοποιούνται πολύ περιορισμένα από τις ε, δυνάμεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Όχι τόσο γρήγορα μου λένε, λέει ο Μιλήτρια. Ζητώ συγγνώμη, νόμιζα ότι με πίεζε ο χρόνος, λέει ο Μιλήτρια, να μιλάω πιο αργά. Ευχαριστούν οι διερμηνείς. Το πρόβλημα λοιπόν έλεγα είναι μια έλλειψη εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα της Ιταλικής κοινωνίας προκειμένου να αναγνωρίζεται η οικογενειακή βία που συχνά μπερδεύεται με την απλή οικογενειακή διαφωνία η οποία διαφορά δηλαδή, η οποία θα μπορούσε να διέπεται από κάποια ε, διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ακόμα. Μόνο 13 από τις 100 νομαρχίες στη χώρα μας, διευρυμένες νομαρχίες, εφαρμόζουν το σχετικό αυτό μέτρο, παρότι γνωρίζουμε ότι η δικτύωση μεταξύ των κέντρων κατά της βίας και των αστυνομικών και άλλων κρατικών υπηρεσιών είναι απολύτως θεμελιώδου σημασίας. Η αμλήτρια δεν έχει επιβραδύνει καθόλου. Μαζί με την υλοποίηση λοιπόν του προγράμματος HELP είναι πολύ σημαντική η συνεχιζόμενη κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων, των αστυνομικών, των διδασκόντων, των ιατρών, των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα έχουν το καθήκον να προστατεύσουν, να υποδεχθούν, να προσφέρουν καταφύγιο στα θύματα και να αναγνωρίσουν τα κρούσματα βίας μεταξύ των φίλων και οικογενειακής βίας. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους την νεολαία μας στα σχολεία προκειμένου να κατανοήσει ότι όταν δεν υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη, στοργή. Και μαζί με τους πόρους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό, θα έλεγα ότι όλες, όλα αυτά τα κονδύλια τα έχουμε απολύτως, απολύτως ανάγκη, ιδιαίτερα στον νότο της Ευρώπης. Και προκειμένου να αλλάξει κάτι διαρθρωτικά είναι απαραίτητη η συνεισφορά των πανεπιστημίων, ώστε σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μαζί με την κατάρτιση όλων των λειτουργών που ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία εκείνα της κατάρτισης που θα βοηθούν όλους αυτούς τους λειτουργούς να αναγνωρίζουν τα φαινόμενα και να διαχειρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο αυτά τα κρούσματα και να λαμβάνουν σωστές και δίκαιες αποφάσεις. Ήδη από τη φάση της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επομένως, όχι μόνο η επικύρωση είναι σημαντική της συμβάσεως, αλλά και η αποτελεσματική εφαρμογή της. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί πολλά ακόμα να συνεισφέρει προκειμένου να προωθήσει μια οδηγία για τα κρατημέλη προκειμένου να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την οδό αυτή, την κατεύθυνση αυτή με αποφασιστικότητα. Υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας. Μια διπλή θυματοποίηση ακριβώς επειδή δεν διακρίνουμε μεταξύ οικογενειακής βίας και διαφορών μεταξύ των συντρόφων ευρύτερα, την ώρα που γίνεται η οποιαδήποτε καταγγελία και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα, να εξεταστούν μάλλον η ποινική διαδικασία και η αστική διαδικασία για οποιασδήποτε αποφάσεις σχετικά με την ευθύνη για τα παιδιά κτλ. Πολύ συχνά όλα αυτά αντιμετωπίζονται υπό το ίδιο πρίσμα, δεν διαχωρίζονται τα φαινόμενα, δεν τους δίνεται διαφορετικό ειδικό βάρος και ακόμα λαμβάνονται αποφάσεις για τα παιδιά πολύ συχνά δίνοντας για παράδειγμα σε μια οικογένεια με δύο παιδιά ένα τέκνο στην ευθύνη του καθενός παρότι έχει υπάρξει στην περίπτωση εκεί οικογενεια... Ε, κρούσμα οικογενειακής βίας. Νομίζω ότι αυτό είναι άλλο ένα από τα θέματα εκείνα που θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί για να προαγάγουμε ένα σωστό δικαστικό σύστημα που θα πρέπει να προστατεύει και τις γυναίκε και τα παιδιά τους από αυτά τα κρούσματα βίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Κουνσουέλα Ροτρίκε, προέδρο ε, της Επιτροπή Ισότητα του Ισπανικού Κογκρέσου. Σα ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σε αυτήν την αίθουσα εκπροσώπηση ε, όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω ότι όπως θα γνωρίζετε και εμείς στη χώρα μας είχαμε αναπτύξει ένα πρωτοποριακό θα έλεγα νομοθετικό πλαίσιο στην αρχή αυτής της πορείας ε, και ο νομοθέτης προσπαθεί να καλύψει εκείνα τα αιτήματα, εκείνες τις ανάγκες της κοινωνίας που καταγράφονται ως υποχρέωση προκειμένου να εξασφαλίσει θεμελιώδη δικαιώματα και να τα προστατεύει. Τώρα για την καταπολέμηση, την ε, Τη οικογενειακή βία και την εξασφάλιση τη ισότητα μεταξύ των φύλων, ο νομοθέτης θα πρέπει να είναι πρωτοπόρο. Παρότι μπορεί η συγκεκριμένη κοινωνία να μην, είναι, να μην είναι έτοιμη να αναλάβει, να εφαρμόσει, να αποδεχθεί πλήρω αυτά τα μέτρα. Μα χρειάζεται το πέρασμα το νομοθετικό προκειμένου να επιτύχουμε μια πιο δίκαιη και σωστή κοινωνία. Αυτό συνέβη και στην Ισπανία. Πέρασαν τα χρόνια, πέρασε ο καιρό και αντιμετωπίζουμε μια η πραγματικότητα, τα στοιχεία μας λένε ότι δεν κάνουμε, αυτά που κάνουμε δεν είναι αρκετά. Αυτά που κάνουμε δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν με τα κρούσματα βίας που είναι μια απόλυτη μάστη αυτή τη στιγμή. Και δεν φτάνει να κρατούμε ενός λεπτού σιγή ή συμβολικά να εκφράζουμε τη λύπη μας ή την αγανάκτησή μας το νομοθετικό πλαίσιο, οι διεθνείς συμφωνίες χωρίς πολιτική βούληση δεν θα χρησιμεύσουν σε τίποτα. Και μάλιστα εγώ θα έλεγα όχι μόνο η πολιτική βούληση αλλά και η δημοσιονομική στήριξη γιατί στην πράξη αυτό σημαίνει υλοποίηση. Και σε αυτό το πλαίσιο στην Επιτροπή Ισότητας της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω υπό την Ισπανική γερουσία, αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο είναι να αντιμετωπίσουμε τα δραματικά αυτά φαινόμενα βίβαιας και γι' αυτό προχωρήσαμε σε ένα σύμφωνο, κρατικό σύμφωνο στο Εθνικό Κοινοβούλιο το οποίο συνυπέγραψαν όλες οι πολιτικές ομάδες της Βουλής. και αυτό που είναι αρκετά προβλέψιμο είναι ότι αν κάθε πολιτική ομάδα ε, διαπραγματευόταν από πλευρά τη από μόνη τη το σύμφωνο, θα είχαμε κατελέξει κάτι τελείω διαφορετικό και αυτό συχνά το τονίζουν και τα μέσα ενημέρωση. Πρέπει να είμαστε ικανοί να παραμερίζουμε το ιδιαίτερο ή στενό κομματικό μας συμφέρον για να επιτύχουμε ένα σύμφωνο το οποίο θα μπορούν να προσυπογράφουν όλοι, το οποίο και επιτύχαμε μέχρι εκείνο το βαθμό. Και το σύμφωνο αυτό έχει δύο βασικούς άξονες και μεθολογία εργασίας. Έχουμε καταρχάς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ισότητα των φύλων, εκπρόσωπους ε, ε, κρατικών υπηρεσιών και φορέων, δικαστικών ε, λειτουργών, φεμινιστικών ενώσεων και για μια ακόμα φορά έχω να ευχαριστήσω θερμά όλες αυτές τι ενώσει γιατί δεν θα είχαμε φτάσει εδώ χωρίς τη δική τους υποστήριξη και το δικό τους αγώνα. Και από την άλλη, συμπληρώνοντας αυτές τις ακροάσεις ε, εμπειρογνωμόνων, αυτή τη δουλειά των εμπειρογνωμόνων, με τη δουλειά των πολιτικών ομάδων. Την κοινοβουλευτική τους δηλαδή δουλειά. Έχουμε τρία τμήματα στο σύμφωνο αυτό το πρώτο τμήμα αναφέρεται σε μια διάγνωση, μια ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης, γιατί βεβαίως για να προκειμένου να κάνουμε σε ένα σύμφωνο πρέπει προηγουμένω να έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας να έχουμε δει τι δεν λειτουργεί καλά, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Την καλή λειτουργία των δημοσίων φορέων και δημοσίων αρχών που πρέπει να παρέχουν το απαραίτητο πλαίσιο ώστε να μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία ισότιμη μια κοινωνία που θεωρεί τον εαυτό της δημοκρατική δεν μπορεί να ε, εξακολουθεί να ανέχεται τα δραματικά φαινόμενα που καταγράφονται αυτή τη στιγμή και που τα υφίστανται οι γυναίκες, αλλά όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και τα ανήλικα συχνά παιδιά τους. Γιατί αυτά ακριβώς τα παιδιά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά ως μοχλός εκβιασμού από πλευρά των δραστών, αυτών που είναι υπεύθυνοι για την άσκηση αυτής της βίας. Δεν μπορεί λοιπόν μια κοινωνία που ισχυρίζεται ότι στον 21ο αιώνα είναι μια προχωρημένη κοινωνία να εξακολουθήσει να ανοίγεται αυτά τα φαινόμενα. Και δεν χρειάζεται απλώς να σημειώνει ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα αλλά να λάβει δράση. Όλες λοιπόν οι διατάξεις 213 στο σύνολο στο ε, σύμφωνα αυτό προκειμένου να λάβουμε δράση. Έχουμε ευαισθητοποίηση, καλύτερη ενημέρωση, ε, θεσμικές ε, απαντήσεις, προστασία των θυμάτων, προστασία των ανηλίκων, κατάρτιση των διαφόρων κρατικών λειτουργών που παρεμβαίνουν σε όλη την αλυσίδα αυτής της διαδικασίας από την καταγγελία μέχρι τη δίωξη, συστάσεις προς τις δημόσιες αρχές και αρμόδιους κρατικούς φορείς και η οικονομική δέσμευση που αναλαμβάνει το σύμφωνο αυτό, δημοσιονομική δηλαδή στήριξη, για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Τώρα, καθένα από αυτά τα 213 μέτρα δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει από κοινού να λειτουργήσουν, αλλά είναι όλα απαραίτητα. Αυτή η συμφωνία υποστηρίζεται και από ένα δισεκατομμύριο συνολικά ευρώ για τα επόμενα πέντε έτη από πλευρά του κράτους αλλά από πλευρά και των αυτόνομων περιφερειών και των δήμων με τη δέσμευση ότι αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα ήδη υπό τον προϋπολογισμό του φετινό. Και θα ήθελα να σχολιάσω το εξή. Τα κρούσματα αυτά βίας Ε, σημαίνουν ενοχικά σύνδρομα, σημαίνουν ταλαιπωρία, σημαίνουν τρόμο, αλλά πάνω απ' όλα σημαίνουν σιωπή. Πολύ συχνά σιγή του θύματος που αισθάνεται ότι απειλείται, σιωπή ε, της ευρύτερης ε, οικογένειας, των φίλων, της κοινωνίας τελικώς. Απέναντι σε φαινόμενα για τα οποία θα έπρεπε να κραυγάζουμε και όχι να σιωπούμε. Επομένως για να μπορέσουμε να συντρίψουμε το, τα τείχη αυτά που έχουν υψωθεί από το φόβο, από τον τρόμο, θα πρέπει να επιμείνουμε. Και από τότε που έχουμε στη διάθεσή μας στατιστικά δεδομένα για τα, κρέμα, για τα κρούσματα βίας αυτά, έχουμε τόσα θύματα σχεδόν όσα και υπό την, ε, τις τρομοκρατικές επιθέσεις ΕΤΑ. Έχουμε οκτώ ανήλικα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Έχουμε τα ίδια μεγέθη Έχουμε τον ίδιο ε, ε, αριθμό φόνων κατά γυναικών ε, στα έτος 16 όπως και στο 15 και έχουμε περί 140.000 καταγγελίες το 16. και πάνω το 80% των γυναικών που υφίστανται κακοποίηση γνωρίζουμε ότι δεν το καταγγέλουν. Επομένως, πολύ συχνά είναι, είναι αρκετά παράδοξο περίεργο να ακούει κανείς ε, για ψευδείς καταγγελίες. Και παραπέμπω και στην ε, δήλωση της ε, συναδέλφου από την περιφέρεια των Βάσκων Γιατί από ό,τι φαίνεται σε εκείνο το κρούσμα της επίθεσης 5 ανδρών κατά της 18χρονης η άμεση, ο άμεσος περίγυρος τοποθετήθηκε υπέρ των 5 και όχι της ε, νεαρής. Τώρα βέβαια εγώ εδώ εκπροσωπώ την, το Ισπανικό Κοινοβούλιο αλλά είναι η ίδια η κοινωνία που θα πρέπει να υποστηρίζει μια τέτοια νεαρή η οποία το βασικό της αδίκημα είναι ότι κατάφερε να επιβιώσει τελικώς. Γι' αυτό κατηγορείται, ότι κατάφερε να επιβιώσει και να συνεχίσει τη ζωή της. Και έχουμε και οπισθοχωρήσει σε σχέση με την ερμηνεία που έχουμε αυτή τη στιγμή των φαινομένων βίας, γιατί πολύ συχνά έχουμε σεξιστικές ερμηνείες που υπερισχύουν, έτσι παλαιού τύπου ρομαντικές, ως έκφραση αγάπης δήθεν. Ενώ είναι απλά και στιγνά κρούσματα βίας. Αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και για να κλείσω να πω απλώς ότι θα συνεχίσουμε όλοι οι δημόσιοι φορές και ιδιαίτερα οι νομοθέτες να κάνουμε τη δουλειά που μπορούμε για να σπάσουμε τη συγκία αυτή, για να παρακάμψουμε την τρομοκρατία και για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Ροντρίγκες. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Ζάκη Αντ, ε, διευθύντρια του Equality Now. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή συνεδρίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλώ σε νομοθέτες ε, όταν προσπαθούμε να επιτύχουμε την εφαρμογή της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Το Εκόλυτο ΝΑΟ ε, είναι ένα διεθνές δίκτυο, προσπαθεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών και χρησιμοποιούμε ως μέσο την νομοθεσία ε, περιφερειακές και διεθνείς συνθήκες που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που δεν τα καταφέρνουμε όμως να κάνουμε είναι να δαμάσουμε την τεχνολογία. Τέλος πάντων, ε, κάναμε μια επισκόπηση της νομοθεσίας για τη σεξουαλική βία. Ε, καλύψαμε 82 χώρες, ε, μεταξύ των οποίων και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο κάναμε την αναθεώρηση αυτή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας εξηγήσω. Γνωρίζουμε την κλίμακα της βίας κατά των γυναικών, κυρίως σεξουαλική βία ε, και κυρίως ε, ε, μετά την εκστρατεία μας όλοι πλέον γνωρίζουν για τη σεξουαλική βία σε όλο τον κόσμο και πόσες, χώρες, πόσες γυναίκες συγγνώμη, πλήττονται από αυτή. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρξαν πάρα πολλά κενά προστασία των γυναικών στην νομοθεσία. Ξέρουμε ότι ο νόμο δεν είναι απάντηση σε όλα. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε αλλαγέ στην νοοτροπία, χρειαζόμαστε εκπαίδευση, χρειαζόμαστε εφαρμογή του νόμου, αλλά ένα, το οποίο, ένα από τα πράγματα που θα έπρεπε να εξετάσουμε πρώτα, πιστεύουμε ότι είναι κάνει τη δουλειά του ο νόμο όσον αφορά την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών. Είδαμε επτά ε, κενά τα οποία θεωρούμε ότι ίσχυαν σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τις ε, διατρέξω εντάχει. Υπάρχουν νόμοι που δίνουν τη δυνατότητα, υπάρχουν νόμοι που δίνουν τη δυνατότητα στους δράστες να φύγουν μετά από κάποιο διακανονισμό με το θύμα ε, γάμος για παράδειγμα ή χρήματα ή κάτι διαφορετικό. Κάποιος διακανονισμός πάντως. Αυτό που σημαίνει πάντως είναι ότι α, εκείνος δεν τιμωρείται και εκείνη δεν δικαιώνεται. Επίσης ε, υπάρχει πολλές φορές μία βάση ηθικής ε, αντί ε, της σωματικής ακεραιότητας και πολλές φορές εξετάζουμε αυτό και δεν εξετάζουμε τη βία που ασκείται πάνω στη γυναίκα. Για παράδειγμα υπάρχουν κάποιοι νόμοι που καλύπτουν το γεγονός ότι υπάρχει βιασμός και στο πλαίσιο της οικογένειας, καμιά φορά και των παιδιών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει, να μην συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην Ινδία οποία υπήρξε μία απόφαση δικαστηρίου που λέει ότι εντάξει αν η νύφη σου είναι πάνω από 15 χρονών μπορείς να τη βιάσεις στο πλαίσιο ενός γάμου. Υπάρχουν διάφορες πρακτικές ε, που δίνουν τη δυνατότητα, στου, τη διακριτική ευκαιρία σε δικαστές ε, να θεωρήσουν ότι κάποια αποδεικτικά ε, συστήματα ε, ε, αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ε, ότι οι γυναίκες δεν είναι θύματα ε, ή ας πούμε το βλέπουμε αυτό σε σχέση με ε, ανήλικα ε, έφηβα κορίτσια τα οποία θεωρούν ότι δελεάζουν τους άντρες, τους προκαλούν και είναι κάτι το οποίο σε μερικά νομοθετικά συστήματα θεωρείται κάποιο ελαφρυντικό. Βλέπουμε ότι, υπάρχει, ότι είναι πολύ ευάλωτα τα κορίτσια και οι γυναίκες πολλές φορές και σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα τεράστιο κενό σεβασμού και προστασίας των έφηβων κοριτσιών από τη σεξουαλική βία. Υπάρχουν πρακτικές και νόμοι παρεμπόδισης της δίωξης ε, ε, ή για παράδειγμα παρότρινσης του μάρτυρα αν κάποιος μπορεί να ε, πάει σε έναν γιατρό ο δεν είναι διαθέσιμος στην περιοχή σου όμως πρέπει να πας σε έναν γιατρό για να αποδείξεις ότι έχεις ε, υποστεί βιασμό. Ε, όταν λοιπόν αυτός ο γιατρός δεν ε, υφίσταται, τότε δεν μπορεί κανείς να αποδείξει τίποτα πιστεύουμε ότι η νομοθεσία όντως μετράει, πρέπει οπωσδήποτε να εστιάσουμε στο δράστη. Εκεί πρέπει να γίνεται η εστίαση και εκεί που είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης, δεν μιλάει μόνο για συνένεση, αλλά συνένεση που, γίνεται, ε, που δίδεται εθελοντικά, ε, κατόπιν ελεύθερης βούλησης ενός ανθρώπου και αξιολογείται στο πλαίσιο κάποιων συγκεκριμένων συνθήκων. Ε, όπως είπα και προηγουμένως, βρήκαμε τους τρόπους αυτούς ε, πλαισίωσης του νόμου. Αν ας πούμε ο νόμος βασίζεται στην ηθική, ε, στην τα δικαιώματα των ανδρών, στο σώμα των γυναικών, αν για παράδειγμα ένας βιαστής δεν τιμωρείται καταλήγοντας σε κάποιο συμβιβασμό, δίνει τη αυτό, αυτό δίνει τη... επιτρέπει η ζωή της γυναίκας να ορίζεται από άλλους δηλαδή διαιωνίζεται η βία των δραστών έναντι της γυναίκας και δεν τιμωρείται και δημιουργείται ένα περιβάλλον στο νομικό ε, πλαίσιο σου ε, που ε, είναι ένα περιβάλλον ελέγχου και υποβιβασμού της γυναίκας, ότι η γυναίκα δηλαδή υπόκειται στον άντρα, οπότε υπάρχει ε, επιτρέπεται αυτό σε μερικές χώρες. Ε, υπάρχει ας πούμε εξαίρεση εξαναγκαστικών γάμων ε, ή εγκλημάτων τιμής σε ορισμένες χώρες. Και ο τρόπος διαμόρφωσης των νόμων επιτρέπει στον κόσμο να σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι και Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει σεξουαλική βία υπό ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Πώς είναι δυνατόν ε, να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους περιστατικά στην καθημερινή μας ζωή. Ε, μερικές φορές ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να, για παράδειγμα υπάρχουν νόμοι που πρέπει να σου δείξει, να, να, να, δείξει κάποια γυναίκα ότι ε, πέρα από το βιασμό υπάρχει και επιπλέον σεξουαλική βία. Δηλαδή ο βιασμός δεν φτάνει. Τι πρέπει να έχει κανείς ας πούμε κάποια σημάδια, μόλοπες. Αν δεν υπάρχουν μόλοπες, τι σημαίνει ότι δεν αντισταθηκε Και αυτό τι σημαίνει ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συνενετική. Πολλές φορές δηλαδή ε, οι νόμοι οι ίδιοι ε, δημιουργούν το βάρο στη γυναίκα να αποδείξει πάρα πολλά πράγματα ώστε να αποδείξει ότι υπέστη βία. Ε, πολλοί λένε ότι η νομοθεσία ήταν ε, αποτέλεσμα των, της ανδρικής ειδονής. Ε, πώς όμως ε, ε μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, να ε, αλλάξουμε αυτή την οτροπία ότι όλα είναι ειδωμένα από την οπτική γωνία ε, του άνδρα ε, και από, το, από τις δικές του ανάγκες, από την οπτική γωνία των δικών, τους, των δικών του αναγκών. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε όταν εξετάζουμε τους νόμους αυτούς και ελπίζουμε ότι και εσείς όταν εξετάζετε νέους νόμους ε, κατά της βίας, ε, κατά των γυναικών, πρέπει να υπάρχει εστίαση στο δράστη. Δεν είναι η γυναίκα κατά πόσο έδωσε τη συνένεσή της, είναι ο δράστης ο οποίος ε, προέβη σε εξαναγκασμό. Πρέπει λοιπόν να διαμορφώσετε διαφορετικό τρόπο σκέψης. Η εστίαση να είναι στο δράστη και όχι στο θύμα. Να είναι η δική του ευθύνη και όχι η δική τη. Αυτό θέλουμε να ισχύει για όλους τους νόμους, όχι μόνο για τη σεξουαλική βία, αλλά και για άλλες μορφές βίας ε, τι οποίε υφίσταται η γυναίκα. Να ολοκληρώσω, ε, η σύμβαση του Κωνσταντινούπολη μιλά για τη σεξουαλική διάκριση και αυτό είναι η ρίζα αυτού του οποίου συζητούμε. Θέλουμε να ε, το υπερβούμε αυτό και θέλουμε να εστιάσουμε και πάλι στους δράστες, να περάσουμε από την εστίαση στο, θήκη, θύμα, ε, αλλά στο θήτη, να μην θεωρείται η γυναίκα δηλαδή υποκείμενη στον άνδρα. Τελευταία μου διαφάνεια είναι μια έκκληση όπως βλέπετε, μια έκκληση ε, στα κράτη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την υποστηρίξουν. Ε, θα θέλαμε την κατάργηση κάθε πρακτικής και νόμου που συνιστούν διάκριση κατά των γυναικών, μεταξύ των οποίων ο ορισμός για τη σεξουαλική επίθεση ε, ε, όταν κάτι γίνεται δηλαδή με εξαναγκασμό χωρίς ελεύθερη βούληση θέλουμε οι γυναίκες να έχουν ε, πρόσβαση σε κέντρα που διευκολύνουν την ε, αποκατάσταση των, των τραυμάτων τους θέλουμε οι γυναίκες να μπορούν να πούν τι του συνέβη να μπορέσουν να συνέλθουν από αυτό και θέλουμε να έχουμε μια διατομιακή προσέγγιση να δούμε δηλαδή και τα θέματα της φυλής και τα θέματα των αναπηριών και να υπάρξει κάλυψη των αναγκών αναγκών όλων, κάθε είδους αναγκών. Θέλουμε κάθε χώρα να έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης, πλήρως χρηματοδοτούμενο, ώστε η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να είναι ένα ζωντανό ε, κείμενο, να μπορούμε συνεχώς να εστιάζουμε σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει μια στρατηγική για την βία κατά των γυναικών και να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επικεντρωθεί σε αυτά τα θέματα ώστε η σύμβαση της, Κωνσταντινούπολη Κωνσταντινούπολης ε, να τύχει ε, πλήρους εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τις ομιλήτριες. Ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε σε αυτό το δεύτερο γύρο. Έχουμε, ε, όπως είπαμε, και από το Ευρωκοινοβούλιο, όπως και από το ε, Εθνικά Κοινοβούλιο Μιλητές. Η κυρία Κοσλόφσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές και τις ομιλήτριες γιατί πραγματι... την συγκεκριμένη προηγούμενη ομιλήτρια διότι μίλησε για τις διακρίσεις που γίνονται στην Ισπανία και για την πολιτική που υπάρχει εκεί για την πάταξη αυτού του φαινομένου. Όλη η Ευρώπη κοιτάει προς την Ισπανία και νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε από εσά. Νομίζω ότι η εφαρμογή βέβαια είναι πολύ πιο ε, σκληρή και δύσκολη από τις δηλώσει. Θα πρέπει όλοι μας ως ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυρώσουμε τη σύμβαση, όμως η εφαρμογή είναι το δύσκολο κομμάτι και το πιο σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να συνταχθώ με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που μίλησαν για τη βία. Ας δούμε λίγο τα πράγματα ε, όπως έχουν. Καταρχάς έχουμε μόνο γυναίκες. Εδώ είμαστε και συζητούμε την κατάσταση των θυμάτων, την προστασία τους, ε, τη βοήθεια που μπορούμε να παρέχουμε. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν έχει να κάνει με τα θύματα, όχι με τους θύτες. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης έχει συγκεκριμένα άρθρα, τα οποία αντίστοιχα μιλούν για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και ε, όσον αφορά τους άνδρες σε αυτή την ε, πολιτική κατά της βίας, είναι λίγα τα χρόνια που μπορούμε πλέον να μιλάμε για βία κατά των γυναικών και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα πάνω σε αυτά που είπε και η συνάδελφος Πετρόφσκα. Στην ε, Πολωνία προσπαθήσαμε να περάσουμε αυτό το νόμο που έχουμε τώρα, ένα εθνικό πρόγραμμα που υφίσταται και σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν συνεχώς τροποποιήσεις διαρκώς. Το 2010 άλλαξε όλη η νομοθεσία για τη βία και εισήχθη νέα νομοθεσία στην οποία λέει ότι πλέον είναι ο θήτης αυτός που θα πρέπει να φύγει και όχι το θύμα από το σπίτι. Εδώ, ε, μετά τη συνθήκη, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, έχουμε πια ορίσει το τέλος ε, του, ε, των βιασμών. Δηλαδή, έχουμε εισαγάγει και άλλες μορφές βίας, την βία στο διαδίκτυο δηλαδή. Έχουμε κάνει τα πάντα για να τα περάσουμε όλα αυτά, αλλά από τότε που πέρασε η σύμβαση, από το 2015 είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Υπήρχαν άνθρωποι που ε, έλεγαν να βγούμε από τη σύμβαση. Τουλάχιστον αυτό είπαν οι άνθρωποι από το κόμμα της, ε, του νόμου και της δικαιοσύνης. Χαίρομαι που η κυβέρνηση και εδώ οι εκπρόσωπος είπαν ότι δεν θα βγούμε από τη σύμβαση, θα είστε οι μάρτυρές μας. Την ακούσατε και ελπίζουμε να είπε την αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αγνιέσκα Κοβλόσκα Μανιέβιτς. Και τώρα έχουμε ε, την εκπρόσωπο του τον εκπρόσωπο του Νορβηγικού Κοινοβουλίου που, μας, ε, που θα μας μιλήσει. Ευχαριστώ. Είμαι ο εκπρόσωπος του Νορβηγικού Κοινοβουλίου. Να σας πω ότι το καλοκαίρι εγκρίναμε τη σύμβαση. Πέρασε πολύ ομαλά από το Κοινοβούλιο. Και ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι δεν ήταν για μας πολύ αντιφατική, στην κοινωνία μας τουλάχιστον, αυτή η σύμβαση, ούτε για τους πολιτικούς μας. Είχαμε ήδη καλύψει πολλούς από τους μηχανισμούς που έχει η σύμβαση στην υφιστάμενη νομοθεσία μας. Παρόλα αυτά, τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, κάνοντας την έρευνά μας για την ενδοοικογενειακή βία, είδαμε και διαπιστώσαμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα σε αυτό το διάστημα παρά τους μηχανισμούς, παρά τα μέτρα, τα νούμερα δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουν μειωθεί. Πρέπει μάλλον να έχουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα και αυτό πρέπει να γίνει και στην Νορβηγία που είναι μια φιλελεύθερη χώρα και μια χώρα η οποία έχει μεγάλη θέληση να ε, υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση. Και στην Νορβηγία λοιπόν πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να δώσουμε περισσότερα χρήματα, να επικεντρωθούμε περισσότερο στην έρευνα, περισσότερα χρήματα στην έβρεση μαρτύρων και φυσικά χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις για να είμαστε πιο στοχευμένοι. Νομίζω ότι ότι η σύμβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική βέβαια, διότι θέτει το, στο επίκεντρο το θήτη και αλλάζει ε, το επίκεντρο. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για ανθρώπινα δικαιώματα. Φεύγουμε από τη σκηνή του εγκλήματος. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οπότε μπορούμε να έχουμε ακόμη πιο ισχυρά εργαλεία. Μπορούμε να έχουμε διεθνείς πιέσεις, να έχουμε μάχη ε, ε, αντίστοιχη με αυτή που είχαμε για τη θανατική ποινή, το βασανισμό και τις δικτατορίες. Από τη διεθνή λοιπόν δραστηριοποίηση επιθεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούμε να πάρουμε μαθήματα και για τη βία κατά των γενικών. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και έχουμε και ένα νέο εργαλείο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε όλες τις χώρες μας και στην Νορβηγία μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Γκαρθία από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τα μέλη του πάνελ για τις παρουσιάσεις τους που μας βοηθούν να κάνουμε μια ακτινογραφία σχετικά με την πρόοδο στις διάφορες ε, χώρες μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των κρουσμάτων αυτών. Μπορούμε πλέον να μιλούμε για διάφορε θετικέ πρωτοβουλίε μεταξύ των οποίων είναι και αυτή η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη που είναι ένα δείγμα τη δέσμευση ε, τη πολιτική που υπάρχει, που εκφράζεται πλέον για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί συμφωνούμε όλοι ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μάστιγα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Πολλέ γυναίκε δολοφονούνται απλώ και μόνο λόγω του γεγονότο ότι είναι γυναίκε. Αυτό απαιτεί δέσμευση, απαιτεί προσπάθεια και πρέπει να καταβάλουμε ακόμα πιο έντονε ε, πλέον προσπάθειε ώστε στα διάφορα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσουμε και να παρακολουθήσουμε τα θέματα αυτά και χρειαζόμαστε όπως είπαν και κάποια άλλη μέλη μια οδηγία σχετικά με το θέμα αυτό. Είναι κάτι που διεκδικούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή της θητείας μας, διότι είναι θεμελιώδου σημασίας. Είναι θεμελιώδου σημασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει σχετικά με το θέμα αυτό. Και να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους το θέμα της αρμοδιότητος ή όχι, όπως λέγεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να νομοθετήσει. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που υπήρξε η πολιτική βούληση και που επομένως νομοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις αμφιβολίες. Εδώ πρέπει να γίνει το ίδιο. Πρέπει να έχουμε έναν ορισμό αντίστοιχο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης του τι είναι θύμα, του πώς ορίζεται το κρούσμα, η επίθεση, για να έχουμε κοινέ πολιτικές, για να έχουμε κοινέ διατάξεις νόμου. Γιατί σε μια χώρα μιλούμε για θύμα οικογενειακής βίας, σε άλλη χώρα μιλούμε για απλώς θύμα βίας ή παρενόχλησης. Χρειάζεται λοιπόν μια κάποια εναρμόνιση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ένα συντονισμός των ορισμών αυτών, των διατάξεων αυτών. Με τη συνεργασία των εκπροσωπών των Εθνικών Κοινοβουλίων, ώστε να έχουμε ακόμα πιο έντιμο, ε, έντονο με συγχωρείτε, το αίτημα αυτό προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρόταση νομοθεσία. Διότι συμφωνώ απολύτω με την Πιλάρ που εκπροσωπεί το Ισπανικό Κοινοβούλιο ότι χωρίς, ότι οι νόμοι δεν αρκούν για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο, αλλά χωρί του νόμου δεν μπορούμε καθόλου να προχωρήσουμε. Και όταν θα έχουμε επιτύχει αυτό, θα πρέπει να δούμε τι άλλο μα λείπει για να συνεχίσουμε την προσπάθεια στις κοινωνίες μας για να ζητούμε και τα υπόλοιπα μέσα που μας χρειάζεται προκειμένου να έχουμε πρόοδο. Χωρίς όμως την νομοθετική πρόοδο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι από εμά εξαρτάται να πολεμήσουμε για μια κοινωνία που σήμερα δεν είναι δίκαιη, δεν, είναι, δεν αντιμετωπίζει τα μέλη της ισότιμα για να έχουμε να γίνουν πραγματικότητα αυτές οι πολιτικές υπό την έννοια της δικαιοσύνης και τη ισότιμη μεταχείρισης όσου κεντρικέ αρχές Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να ενώσετε τις φωνές σας μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλζα Πάης από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς δεν ακούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι η χώρα μου ήταν η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επικύρωσε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το 2013. Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοκογενειακής βίας ε, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης Πορτογαλία. Υπήρξαν καταγγελίες ε, ε, και πολλές πολλά προβλήματα στην καταγραφή αυτών των ε, καταγγελιών. Ε, ε, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες κάθε χρόνο στα αστυνομικά τμήματα. 20 άτομα δολοφονήθηκαν από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους πέρσι στην Πορτογαλία. Ε, και νομίζω ότι επειδή γίνονται πια γνωστά αυτά, ε, επειδή είναι γενναία πια τα θύματα και ε, καταγγέλουν την κατάσταση αυτή, είναι, η σιωπή αυτή σταματά να υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο η ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει και ο ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων και άλλου είδους βία που αφορά τα άτομα ε, ΛΟΑΤ επίσης ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η απάντηση να δοθεί ε, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το κάθε θύμα. Το Κοινοβούλιο έχει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής δεν χρειαζόμαστε νόμους για τα πάντα. Υπήρχε όμως ένας νόμος το 2017 που προέκυψε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των παιδιών σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των γονέων. Η Σύμβαση λέει ότι πρέπει τα παιδιά να προστατεύονται χωρίς ε, να ε, μην υπάρχει προστασία βέβαια για τις μητέρες τους. Οπότε υπήρξε μια, ε, ένας νόμος σε σχέση με τη γονεϊκή ευθύνη όταν τα παιδιά είναι θύματα της βίας, γιατί συνήθως τα πρώτα θύματα είναι τα παιδιά. Θέλουμε και έναν προϋπολογισμό που έχει να κάνει συγκεκριμένα ε, με τα θέματα αυτά των φύλων σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής. Θεωρούμε ότι αυτό ε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο προϋπολογισμός ενδοικογενειακής βίας για την ενδοικογενειακή βία έχει επίσης ενισχυθεί και έχουμε ένα νέο σύστημα που ε, προωθεί ε, την ισότητα ε, στο πλαίσιο των σχολείων. Έχουμε δει λοιπόν ότι τα πάντα μπορούν να... Ε, οι αγώνες μπορούν να δοθούν και σε επίπεδο σχολείου. Δεν υπάρχει μόνο ο νόμος, υπάρχει και η σχολική εκπαίδευση που μπορεί να βοηθήσει. Αν δεν έχουμε το σθένος να μάθουμε αυτά τα πράγματα στα παιδιά από νωρίς και να τους πούμε ότι δεν πρέπει να, είναι, να, να, μπαίνουμε σε δυναστικές σχέσεις ε, όπου κάποιος άλλος είναι ο κυρίαρχος ε, και εμείς τα θύματα, ε, τότε μόνο μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη. Όταν κερδίσουμε τη μάχη για να κερδίσουμε τη μάχη αυτή πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει ισχυρή νομοθεσία και επίσης πρέπει να υπάρξουν νόμοι που θα ενθαρρύνουν τις αλλαγές αυτές. Κύριος Κρίμπεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να... Μάλλον είναι δύο ανοιχτά τα μικρόφωνα στην αίθουσα να κλείσει αυτό που δεν χρησιμοποιείται από τον ομιλητή. Εδώ μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών, των παιδιών, των ε, ηλικιωμένων, όμως ε, το βασικό θέμα είναι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό που μας αφορά κυρίως ε, εδώ, παρόλο που οι γυναίκες είναι στο προσκήνιο, είναι κάτι πολύ αντιφατικό. Πολλά ε, κράτη έχουν πρόβλημα με τη σύμβαση. Ναι, η σύμβαση ασχολείται με τη βία κατά των γυναικών, αλλά βασίζεται κυρίως σε έμφυλη ιδεολογία η οποία είναι αντίθετη με τις αρχές πολλών ανθρώπων μεταξύ άλλων και των συντηρητικών πολιτικών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε πόσο καλό είναι ένα έγγραφο όταν είναι απαράδεκτα πολλά από τα άρθρα του. Η ιδεολογία στην Νορβηγία, για παράδειγμα, ε, ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος έδειξε πόσο γελία ήταν αυτή η ιδεολογία για το φύλλο. Υπάρχουν επίσης έννοιες που έρχονται σε αντιπαράθεση με την εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων και η έννοια του φίλου. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Φοβάμαι ότι εδώ έχουμε παραβίαση των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έγγραφο και η πίεση για την κύρωση στην ουσία διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση Νομίζω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να λύνεται εντός των κρατών μελών, θα πρέπει να υπάρχει προστασία για τα θύματα, να υπάρχουν κάποιες εκστρατείες για την πρόληψη, αλλά δεν πρέπει να κυρώσουμε αυτή τη σύμβαση. Χρειαζόμαστε άλλο έγγραφο, καλύτερο. Η ενδοοικογενειακή βία είναι πραγματικά δραματική και αποκρουστική. Όμως, ο τρόπος να την αντιμετωπίσουμε είναι να επικεντρωθούμε στις σχέσεις αγάπης. Ο κύριος Έιντα μίλησε για 20 χρόνια νομοθέτησης που δεν άλλαξε τα νούμερα. Αυτό είναι μια ιδεολογική προσέγγιση εμείς. Τι χρειαζόμαστε. χρειαζόμαστε μάλλον να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Πολύ συχνά οι δράστες ε, τη γλιτώνουν ε, χάρη σε άλλες νομοθεσίες. Αν ακούσουμε όλους τους ανθρώπους ε, που ε, είναι χριστιανοί, Εβραίοι κτλ. Ε, θα καταλάβουμε ότι δεν θέλουμε αυτή τη φιλετική ιδεολογία. Οι γυναίκες και οι άντρες είναι ίσοι, υπάρχουν πράγματα που οι γυναίκες τα κάνουν καλύτερα ε, και οι άντρες που αγαπούν τις γυναίκες τις φροντίζουν, τέτοια πράγματα. Μέλη Παρλαμέντας Εδώ είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι λίγο έχουμε ε, διάφορες απόψεις, ε, τα πνεύματα λίγο οξύνονται. Ε, έχουμε τώρα και τη Λιθουανία. Είναι και αυτή μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. είμαι καθολική κι εγώ και ε, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη βία κατά των γυναικών σε καμία χώρα, ούτε με τις παραδόσεις, ούτε με τη θρησκεία. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να σταματήσει αυτή η ιδεολογική προσέγγιση. Τώρα πάμε στη Ρουμανία. Από... Κυρία Πρόεδρε, είμαι από τη Ρουμανία, μια ε, χώρα από την κεντρική η Ανατολική Ευρώπη. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και βλέπω πολλές φίλες, στην Τζεραλντίνα, τη Λίζα, πολλές φίλες και φίλους από το δίκτυο κατά της βίας και πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια να πω ότι ότι η Ρουμανία δεν είναι απλώς παρατηρητής, αλλά μια χώρα που έχει προσυπογράψει και κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, έχει εφαρμόσει τη σύμβαση και έχει κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο πρωτογενές και δευτερογενές και τριτογενές δίκαιό της. Δεδομένου του λίγου χρόνου που έχω θα σας δώσω λίγα παραδείγματα. Έχουμε τους περιοριστικούς όρους ε, και υπάρχει μια διαδικασία τροποποίησης της νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 52 της Σύμβασης, ε, η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει. Ε, μιλάμε για όλες τις μορφές παρενόχλησης και την νομοθεσία που ασχολείται με αυτή και για την έμφυλη βία. Αλλά μιλάμε και για την χρηματοδότηση των καταφύγιων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε την νομοθεσία και εγώ σας μιλώ εδώ ως δικηγόρος, όμως ταυτόχρονα ο τρόπος εφαρμογής της νομοθεσίας αποτελεί κλειδί. Ε, είναι κρίσιμο σημείο και θεωρώ ότι ένα απαραίτητο νομικό πλαίσιο θα μας βοηθήσει. Μιλάω και ε, από την πλευρά της δικής μας χώρας όπου κάναμε μεγάλη μάχη ε, και δεν κάναμε υποχωρήσεις για την νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό παρόλα αυτά να ληφθούν τα μέτρα πρόληψης της βίας πριν συμβεί. Και είμαι χαρούμενη που άκουσα και σήμερα να βάζουμε το επίκεντρο, στο επίκεντρο αυτό το θέμα. Οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων και εδώ και στη χώρα μου κάνουν εξαιρετική δουλειά. Πρέπει πάντοτε να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας ε, για τη δουλειά που κάνουν, γιατί πραγματικά η εκπαίδευση και η πρόληψη είναι πολύ σημαντικά βήματα σε αυτή τη μάχη. Είναι ο τρόπος να προβλέψουμε και να ελεγχιστοποιήσουμε τη βία και τις διακρίσεις. Θα συνεχίσω λέγοντας ότι ε, μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία χωρίς βία όπου οι γυναίκες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες και ποτέ δεν είναι αργά. Καλό είναι να απαλλαγούμε από αυτό το παράσιτο στην κοινωνία μας, ε, να ζούμε χωρίς βία, διότι υπάρχουν εκατομμύρια γυναικών ε, που αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ε, πάσχουν, υποφέρουν από τη βία στα χέρια ε, ανθρώπων ε, που και η βία αυτή γίνεται ανεκτή από το κράτος τους. Και γι' αυτό η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εκπροσωπεί μια κοινή πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών χωρών. Ακόμα και με τέτοιες εκδηλώσεις όπως η σημερινή που μαθαίνουμε ένας από τον άλλον, προωθούμε καλές μορφές συνεργασίας. Σας ζητώ λοιπόν να συνταχθείτε μαζί μου και να πούμε όλοι μαζί σήμερα ότι ο βασικός μας στόχος είναι να σταματήσουμε τη βία, γιατί η βία οδηγεί σε βία. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ. Κυρία Βαλινάκη. Κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμένα μου φαίνονται επικίνδυνες κάποιες από τις απόψεις των μελών που εκφράζονται εδώ, λέει ο Μιλήτρια, και εκτός τόπου. Η Ισπανία επικύρωσε τη σύμβαση, ετέθη ενισχύ από την 1η Αυγούστου του 2014. Εγώ πιστεύω ότι η χώρα μάλλον αγνοεί με κάποιο τρόπο την όλη σύμβαση, εκτός αν η δικαστική λειτουργία απλά δεν το διάβασαν, δεν γνωρίζω. Η δικαστική αυτή απόφαση στην οποία αναφέρθηκε η συνάδελφος ε, σχετικά με την επίθεση των πέντε ανδρών, για να τους αποκαλέσω έτσι, βιάζουν μια 18χρονη με δύο αστυνομικούς και έναν στρατιωτικό με προηγούμενες καταδίκες για επιθέσεις βίες κτλ. Όπου το δικαστήριο αρνείται την μελέτη που υποβάλλεται από ιδιωτικό ερευνητή ενός συνδεδεμένου οικογενειακού μέλος αρνείται τις ενδείξεις WhatsApp που είχε, στη, τα μηνύματα δηλαδή, στη διάθεσή του μεταξύ των θητών και που αυτή τη στιγμή στην ουσία ε, το δικαστήριο προχωρεί σε μια ηθική τοποθέτηση, απόφαση, επίκριση κατά του θύματος. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά που λέμε, η σύμβαση και τα υπόλοιπα, να γίνουν πραγματικότητα, γιατί διαφορετικά η ευθύνη των των παιδιών, για παράδειγμα, στο οποίο επίσημα αναφέρει και μια συνάδελφος, που δίδεται συχνά σε ανθρώπους που έχουν διαπράξει ποινικά δικήματα. Χωρίς άλλη επιτήρηση. Όπου έχουμε δολοφονίες, περίπτωση δολοφονίας μπροστά στα παιδιά της, γυναίκας από το σύντροφό της με τέσσερις προηγούμενες καταγγελίες και επιθέσεις. Μπροστά στα παιδιά της και μπροστά στην πόρτα του σχολείου. Θέλω να πω, πιστεύω ότι οι γυναίκες πρέπει να υπερβούμε τις ιδεολογικές, τις κομματικές μάλλον τοποθετήσεις και τουλάχιστον αναφέρομαι στη χώρα μου. Κανένα κόμμα δε, δεν ηγείται από γυναίκα. Υπάρχει ένα πατριαρχικό σύστημα που βασιλεύει απολύτως στη χώρα μας. Στη χώρα μας τουλάχιστον. Για να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πρόκειται για την προστασία των δικαιωμάτων μας και της ισότητας την οποία δικαιούμαστε. Και δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται ακόμα και στα πλαίσια πολιτικών λιτότητος που πλέον ακολουθούμε εκπτώσεις σε αυτά τα θέματα. Γιατί εκεί αμέσως στρέφονται καταρχήν οι κυβερνήσει όταν έχουν να λάβουν μέτρα λιτότητα. Κόβουν οποιαδήποτε βοήθεια από τέτοια κοινωνικά ζητήματα. Στην Ισπανία άνω του 90% των γυναικών που έχουν δολοφονηθεί λέγεται στην Ισπανία, σύμφωνα με μελέτες, ότι δεν είχαν υποστεί σωματική βία, μόνο ψυχολογική προηγουμένω. Δηλαδή αυτό είναι μια ένδειξη τοποθέτηση των δικαστικών λειτουργών, των δικαστηρίων. Γιατί ίσως τελικά αυτό που επιδιώκεται με αε είναι οι γυναίκε να μην καταγγέλουν καν τα επεισόδια αυτά, τα κρούσματα αυτά, τις επιθέσεις που δέχονται. Επομένως πέρα από συμβάσεις χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται κατάρτιση και των δικαστηρίων, των δικαστικών λειτουργών, γιατί βλέπουμε οπισθοδρόμηση πραγματική και σκανδαλώδης τοποθετήσει και αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φραδίτη Σταμπούλη έχει το λόγο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα υπάρχει από το 2006 νομοθεσία η οποία διώκει αυτεπάγγελτα την ενδοοικογενειακή βία η οποία ενδοοικογενειακή βία, για να μην γελιόμαστε, αφορά στη συντριπτική της πλειοψηφία γυναίκες και είναι βία λόγω φύλου. Στη συντριπτική πλειοψηφία, επαναλαμβάνω. Η ίδια νομοθεσία διώκει το βιασμό αντός του γάμου και προβλέπει δωρεάν νομική βοήθεια για τα θύματα και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του δράστη. Υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων λειτουργεί η γραμμή ΣΟΝΣ όλο το 24ωρο και υπάρχουν 40 συμβουλευτικά κέντρα και 21 κέντρα φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους, όπου επίσης παρέχεται συμβουλευτική εργασία. Τα κέντρα αυτά χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο νόμος προβλέπει επίσης διαδικασία ποινική διαμεσολάβησης, η οποία έχει σχετικά περιορισμένη εφαρμογή, αλλά και έχει επισύρει και αρνητικές κριτικές. Επίσης, από το 2017 ενσωματώθηκε στην νομοθεσία μας η Οδηγία 2012-29 Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικότητας χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνότητας, γλώσσας, θρησκείας, κοινωνικής προέλευσης, πολιτικών ή άλλων πεπιθήσεων, περιουσιακής κατάστασης, ηλικία, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λειτουργεί η Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης. Με αυτή την υποδομή λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση προχωρεί στην κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Το σχετικό νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στις 17 Νοεμβρίου για διαβούλευση η οποία λήγει στις 2 Δεκεμβρίου. Άρα το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση αν όχι τι τελευταίε εβδομάδε του 2017 τις πρώτες εβδομάδες του 2018. Και αυτή θεωρώ ότι είναι μια καλή είδηση και είμαι πολύ ευχαριστημένη που είμαι σε θέση να σας την ανακοινώσω σήμερα. Εκτός από την κύρωση της σύμβασης, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αλλαγές στην νομοθεσία ώστε οι διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας να περιλαμβάνουν και τα μέλη του Συμφώνου Συμβίωσης, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία από το 2016 μπορούν να ανήκουν και στο ίδιο φύλλο. Αντιμετωπίζονται θέματα αποζημίωσης των θυμάτων, γιατί η προηγούμενη νομοθεσία έχει ατέλειες. Απαγορεύεται η οπλοφορία στους δράστες ενδοοικογενειακής βίας και απαγορεύεται η επιστροφή αλλοδαπού, αλλοδαπής στην ουσία, θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, θεσμοθετείται όχι μόνο η παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των μορφών βίας που καλύπτει η Σύμβαση, αλλά και η συλλογή αναλυτικών σχετικών στατιστικών στοιχείων κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Μέσα στο 2018 θα πρέπει να επιληθεί το θέμα της χρηματοδότησης των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενικής βίας για το 2019, είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον μάλιστα όπως αναμένεται η χώρα θα έχει βγει από την Επιτροπή και θα μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κοινωνική πολιτική σύμφωνα με τις πεπιθήσεις της, είτε με ανανέωση των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων τόσο για τις χώρες που ήδη έχουν κυρώσει τη σύμβαση, όσο και για εκείνες που θα το κάνουν από τώρα και ύστερα. Βεβαίως όπως είπανε πολλές προλαλήσασες και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, η νομοθεσία είναι αναγκαία, αλλά αναγκαιό, ε, αναμφισβήτητη αναγκαιότητα παραμένει η αμφισβήτηση των στερεοτύπων του φύλου από ένα γυναικείο φεμινιστικό κίνημα που θα ενδυναμώσει τις γυναίκες αποτρέποντας τη θυματοποίησή τους και που θα διαμορφώσει και το κοινό περιδικαίου αίσθημα ως η δικαστική εφαρμογή της νομοθεσίας να έχει τα αποτελέσματα που έχει το πνεύμα του νομοθέτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγιούτο, μέλος Επιτροπής ΦΑΜ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ερχόμενο Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, θα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της ε, βίας κατά των γυναικών. Νομίζω ότι και εγώ και πολλές από τις συνάδελφοι, συναδέλφους με συγχωρείτε, θα, παρουσι... θα κάνουμε σχετικές παρουσιάσεις. Εγώ θα βρίσκομαι σε ένα σχολείο και θα μιλήσω στους ε, μαθητές για να ενθαρρύνω κυρίως τους μαθήτριες να καταγγέλουν τα κρούσματα αυτά βίας. Γιατί το είπαμε, ξεκινάμε με την παιδεία, ξεκινάμε με τα σχολικά συστήματα, αλλά χρειάζεται πολύ θάρρος. Σήμερα, τουλάχιστον στη χώρα μου, για να καταγγείλει κανείς. Το 85% των θυμάτων δεν προχωρούν σε καταγγελία. Γιατί? Διότι τα μέσα που τους δίδονται, που τους παρέχονται, παρότι έχουμε επαρκή νομοθεσία, τα μέσα που τους δίδονται είναι ανεπαρκή για παράδειγμα κατοικίες, χώροι στους οποίους θα μπορούσαν να προστατευτούν αυτά τα θύματα. Και δεν μιλώ κυρίως για τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά για την περιφέρεια, για την επαρχία. Τι κάνουν λοιπόν τα θύματα όταν γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος που μπορεί να τους υποδεχθεί και να τους προστατεύσει. Τίποτα. Σιωπούν. Και υπάρχουν πάρα πολλές ε, συνδεδεμένες αντιδράσεις που μπορούν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την όλη κατάσταση και να οδηγήσουν σε ένα κρούσμα φούνου από εκεί που υπάρχει απλώς αρχικά μία ένταση χωρί και όλα αυτά διότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διαμαρτυρίας επίσημης καταγγελίας. Επομένως η παρακολούθηση που χρειάζεται, αυτή η επιτήρηση την οποία επικαλούμαστε και με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να εγκρίνουμε στα διάφορα εθνικά μας κοινοβούλια σχετικές διατάξεις. Μετά από χρόνια εννοώ. Όμως πλέον έχουμε φτάσει ομόφωνα να εγκρίνουμε σχετικά σχέδια διατάξεων. Επομένως ε, ε, υπάρχει η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση. Ας ε, εξασφαλίσουμε ότι η μη αποτελεσματική υλοποίηση μιας διαταξη δεν θα σημάνει και την αποδυνάμωση τη ίδια της διάταξη υπό την νομική έννοια, υπό την έννοια του δικαίου. Δηλαδή ναι, α νομοθετούμε σωστά και με πληρότητα, αλλά θα πρέπει διαρκώς να ελέγχουμε ότι αυτές οι διατάξεις θα υλοποιούνται και θα προστατεύουν τι γυναίκε. Ε, ε, ε, Ευχαριστούμε κυρία Γιούτα. Η κυρία Περεσνόβα από το Σλοβακικό Κοινοβούλιο. <laughs> Eh, Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε για κάποιες ε, εμπειρίες ε, των γυναικών και γνωρίζω ε, πολλά για γυναίκες θύματα βίας. Για 20 χρόνια έχω βοηθήσει κορίτσια που ήταν θύματα βίας, βίας που υπέστησαν από τους πατέρες τους, για παράδειγμα. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν θα έπρεπε να μας διαχωρίζει Αν δημιουργεί προβλήματα για κάποιες χώρες, τότε για τις γυναίκες και τα κορίτσια που μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ μπορούμε νομίζω να αφήσουμε κατά μέρος τις διαφωνίες μας. Μπορώ να δω και τις δύο πλευρές ε, και τα επιχειρήματά τους. Ε, η Υπουργό Δικαιοσύνης της Σλοβακίας θέλει να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Ε, αν κατάλαβα καλά ε, θέλει να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο σχολών ε, της Σλοβακίας, μίας ε, που θέλει την ταχεία κύρωση και μια ομάδα επιρογνωμόνων που δεν θέλει προσχώρηση στη συγκεκριμένη σύμβαση. Εγώ ανήκω στη δεύτερη σχολή. Θα συνεχίσω να βοηθώ τις γυναίκες θύματα βίας. Το έχω κάνει άλλωστε για 20 χρόνια και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι μιλάω εκ όταν λέω ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δεν είναι ο σωστός τρόπος. Να προχωρήσουμε. Κάποιοι έχουν την προκατάληψη να πιστεύουν ότι όσοι διαφωνούν με τη σύμβαση, διαφωνούν και με την ε, καταπολέμηση της ενδοοικογενειακή βίας. Όχι, εμείς έχουμε νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων βίας 139 ψήφοι υπέρ από τα 145 μέλη που ήταν παρόντα και ψήφισαν ε, η νομοθεσία αυτή προβλέπει την προστασία των θυμάτων μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά και την απαραίτητη χρηματοδότηση για την ε, αντιμετώπιση αυτή. Ασφαλέστερη στέγαση, ε, συμβουλές, ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι σημαντικό να παρέχονται στα θύματα βίας, αλλά το έχουμε αυτό στην εθνική μας νομοθεσία, στη Σλοβακία. Πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε, αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όρτασούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω για τις εισφορές ε, όλων των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι μια συζήτηση, ένας διάλογος που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό σε αυτόν τον Νίκο, σε αυτή την Επιτροπή. Εγώ θεωρώ ότι η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης είναι ένα απολύτως απαραίτητο μέσο. Έχουμε μια κάποια αμφισημία αυτή τη στιγμή σχετικά με την υλοποίησή του, μέσου, της συμβάσεως. Εμείς όμως εργαζόμαστε για να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό και το διεθνέ πλαίσιο είναι απόλυτο απαραίτητο για να μπορέσει να προχωρήσει η εθνική νομοθεσία και θα κράτη μέλη. Αυτό το βλέπω στη χώρα μου αλλά το βλέπω και σε άλλε χώρε. Πολύ συχνά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το Συμβούλιο τη Ευρώπη μα έχουν εξωθήσει, υποχρεώσει τελικά να προχωρήσουμε στην έγκριση δική μας νομοθεσίας. Όμω, αυτή η σύμβαση δεν θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση δικαιολογία για να πούμε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να το δώσουμε ως μήνυμα με αφασιστικό τρόπο στις κυβερνήσεις μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ήταν απαραίτητο να επικυρώσουμε τη σύμβαση, αλλά αυτό δεν είναι κάτι σαν ε, τελικός προορισμό σε καμία περίπτωση. Θέλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να επιτύχουμε και τα υπόλοιπα μέσα που χρειαζόμαστε. Πράγματι νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητη συνθήκη, αλλά δεν είναι και ικανή. Και μιλούμε για ένα πλαίσιο που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, πολύ σκληρό. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί κανείς ε, να χρησιμοποιεί ε, ως ιδεολογία τη διαφορά μεταξύ των φύλων, όπως μερικοί επιχειρούν να κάνουν. Αλλά ήθελα να κλείσω με το εξής σχόλιο. Η βία κατά των γυναικών είναι η ένδειξη μιας αυξανόμενης ανισότητας. Και κάτι από αυτά που έχουμε μπορέσει να δούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χάρη και στην εξαιρετική δουλειά του Ινστιτούτου Ισότητας του Ευρωπαϊκού, όλες, όλοι οι δείκτες ανισότητος μισθολογικής, ε, συνταξιοδοτικής και ό,τι άλλο θέλετε, εάν δεν είναι απλά μπλοκαρισμένοι, δρομούν. Αυτή είναι η γενική τέση. Και το βαθύτερο πρόβλημα είναι ότι στην Ευρώπη έχω την αίσθηση ότι ε, πάμε προς μια ενίσχυση, αναβίωση του πατριαρχικού συστήματος. Μια επιστροφή, δυναμική επιστροφή του πατριαρχικού συστήματος. Και όλα αυτά ενδυναμώνουν και ενθαρρύνουν τα κρούσματα αυτά βίας. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένα μέσα, αλλά αντιμετωπίζοντας τα αίτια που είναι η πραγματική ανισότητα μεταξύ των φίλων, μεταξύ των ανδρών και γυναικών. Και εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ότι το θεματολόγιο της ισότητας έχει φτάσει σε ένα τέλμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι λόγω ελληπού φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή όλε οι σχετικέ πρωτοβουλίε, λέει ο μιλητή, φτάνουν σε ένα τέλμα στο Συμβούλιο τα σχετικά με την άδεια μητρότητα, διάφορες προτάσεις που μπλοκάρονται από το Συμβούλιο. Και καθότι εδώ έχουμε και εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα πρέπει να πιέσετε τα μέλη των εθνικών σας κυβερνήσεως για να προχωρήσουν αυτές οι προτάσεις στο Συμβούλιο. Γιατί το Συμβούλιο τις παγιδεύει και τις μπλοκάρει και μένουν εκεί για πάντα. Είναι απολύτω απαραίτητο για να ξεπεράσουμε αυτό, αυτό το τέλμα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Η κυρία Μπενίτες. ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους ε, υπόλοιπους εκπροσώπους από το Ισπανικό Κοινοβούλιο και από τους υπόλοιπους ισπανικούς φορείς. Νομίζω ότι στη χώρα μας είναι ένα κρατικό θέμα, ένα κρατικό ζήτημα. Και επί τη βάση της νομοθεσίας που εγκρίναμε από το 2013 και μετά, το 2015, έχουμε συμπληρώσει σιγά σιγά το νομοθετικό μας πλαίσιο, τροποποιήθηκαν και οι σχετικές διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων και των τέκνων, από τα κρούσματα βίας. Έχουμε τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα για να αναγνωρίζονται διάφορες, διάφορα δικήματα ε, όπως αναγνωρίζονται και ορίζονται από τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, αλλά με την ευαισθητοποίηση στην οποία έχουμε προχωρήσει στην ισπανική κοινωνία, ε, το 2014 όπως ελέγχθη επικυρώσαμε τη σύμβαση και από τότε έχουμε υλοποιήσει κάποια μέτρα νομοθετικής ανάπτυξης των μέτρων αυτών και ανάπτυξης επίσης στρατηγικής και άλλων πρωτοκόλων που μπορούν να συνοδεύουν αυτές τις πολιτικές. Στο σύμφωνο που εγκρίναμε επίσης ε, ε στην Γερουσία και την Βουλή, ε, στην Ισπανία, Εκπροσωπώντας λοιπόν τη Γερουσία να σας πω ότι το Σεπτέμβριο εγκρίναμε και εμείς, υπερψηφίσαμε αυτό το σύμφωνο που είναι ένα φασιστικό βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και αυτό χάρη στη συνεργασία όλων των πολιτικών κομμάτων της Βουλής ε, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα κομματικό συμφέρον και να μείνουμε στο βασικό άξονα της προστασίας των θυμάτων. Και αυτό χάρη σε μια δέσμευση και πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έθεσε και αυτά, το, αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 5 έτη για όλες τις σχετικές πολιτικές. Να εξηγήσω ότι στη Γερουσία 277 μέτρα έχουν εγκριθεί για όλο το φάσμα των σχετικών αδικημάτων βίας και έχουμε προχωρήσει και στη σχετική τροποποίηση διαφόρων άλλων νομοθετικών πράξεων που χρειάστηκαν στα πλαίσια αυτής της ε, επικαιροποίηση αν θέλετε. Θα έχουμε τη Διεθνή ημέρα για τη βία κατά των γυναικών, η ομιλήτρια μιλάει πάρα πολύ γρήγορα, δεν την προλαβαίνουμε. Το πώς θα λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της προστασίας των ανηλίκων. Μέσω του συμφώνου που έχουμε εγκρίνει, έχουμε εγκρίνει και σημαντικά μέτρα για τους νεαρούς, για τους έφηβους, για τους ανηλίκους, γιατί πρόκειται για μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες σε αυτού του είδους ε, τα κρούσματα Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία συνεχή παρακολούθηση κοινωνικών ε, μέσων δικτύωσης αλλά και κρούσματα βίας που, που το πιο ανησυχητικό είναι ότι ε, γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό μια κοινωνική αποδοχή. Όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα κάνουμε μέσω του συμφώνου που εγκρίναμε για προληπτικά μέτρα μέσω των ε, προγραμμάτων εκπαίδευσης, το είπε και η πρόσωπος της Ιταλικής Γερουσίας. Εστιαζόμενοι βεβαίως στις νέες τεχνολογίες, ξαναλέω, γιατί αυτό είναι ο τρόπος της πιο αποτελεσματικής ευαισθητοποίησης και για να ευαισθητοποιήσουμε τους ε, δασκάλους και τους γονείς, τους κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται με τα παιδιά, τους εκπροσώπους των αστυνομικών δυνάμεων και των δικαστικών λειτουργών, και προχωρούμε σε συνεχείς εξαιρετικές ευαισθητοποίησεις που αφορούν στα παιδιά. όπου εστιαζόμαστε σε αυτόν που διαπράττει το αδίκημα της κακοποίησης ή της βίας. Να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, θέλετε. Απλώς έχουμε εγκρίνει επίσης μια σειρά από μέτρα για να αποφύγουμε την εκμετάλλευση των παιδιών από τους πατέρες ώστε να βλάψουν τις μητέρες τους, λέει ο Σήμερα στην Ισπανία διακόπτεται η... το δικαίωμα της επίσκεψης των πατέρων προς τα παιδιά τους όταν έχουν ε, ληφθεί συγκεκριμένες καταδικαστικές αποφάσεις ή απομάκρυνση από, το... από την αιστεία. Ε, επομένως υπάρχει μια κάποια βελτίωση και ως προς την απόδοση ε, και σχετικά με την ε, ε, υποχρεωτική και η δαιμονία, ε, θέμα στο οποίο αναφέρθηκαν και αρκετοί συνάδελφοι και την οποία παραχωρούν πολύ συχνά τα δικαστήρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το βήμα αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να μας βοηθήσουν στην ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη για να επιτύχουμε μια κοινωνία χωρίς βία και χωρίς βία κατά των γυναικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.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 Sprejeli smo spremembe zakona o preprečevanju nasilja v družini. Να σας πω ότι έχουμε κάνει αλλαγές στον ε, ποινικό μας κώδικα στη Σλοβενία σχετικά με τον πρόωρο και αναγκαστικό γάμο αλλά και με την επίμονη παρακολούθηση μέσω των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, έχουμε επικεντρωθεί στη χρήση των δεδομένων βάσει της συνένεσης. Αλλά έχουμε κάνει και άλλες αλλαγές. Έχουμε εγκρίνει επίσης ε, το ψήφισμα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών. Έχουμε διάφορες προτεραιότητες όπως η μηδενική ενοχή στη βία κατά των γυναικών. Μετά, έχουμε πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες και μέτρα, τα οποία θα δείτε και στο αντίστοιχο ψήφισμα για το Εθνικό Πρόγραμμα σχετικά με την ε, πρόληψη και την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας. Ε, αυτό είναι στη φάση τη σύνταξης και θα το εγκρίνουμε σύντομα. Να ενημερώσω όμως και για κάποια άλλα project που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στη Σλοβενία. Καταρχάς να αναφερθώ στο project Βία κατά των γυναικών, σε ένα άλλο που ονομάζεται «Σταματήστε την ε, επιγραμμική βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλο ένα project που έχει να κάνει με τις ίσες ευκαιρίες ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως και το πρόγραμμα για την πρόληψη της βίας. Έχουμε στατιστικά στοιχεία από την αστυνομία, ε, τα οποία μας βοηθούν στη Σλοβενία. Για την περίοδο μετά την κύρωση της ε, σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Ας πούμε τα πλημελήματα που έχουν και κάποιο στοιχείο ενδοοικογενειακής βίας έχουν μειωθεί, αλλά όχι πάρα πολύ. Απ' την άλλη, τα ποινικά αδικήματα, στα οποία το θύμα είναι γυναίκα, έχουν μειωθεί δραματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, εδώ τελειώνει το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο πάνελ ε, ακούσαμε τους ευρωβουλευτές και ακούσαμε και την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Είναι άλλοι πέντε που ζήτησαν το λόγο, αλλά μάλλον θα μιλήσουν στο τρίτο πάνελ. Θα υπάρχει συζήτηση μετά το τρίτο πάνελ. Να είστε ήσυχοι γι' αυτό. Υπάρχουν τα εθνικά κοινοβούλια που θα μιλήσουν και θα έχουμε και χρόνο για συζήτηση, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο για συζήτηση. Καλό είναι να ακούμε λοιπόν μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και συνάδελφος ε, από την Ισπανία, να ε, ασκήσουμε πίεση και σε όλα τα επίπεδα και στο Συμβούλιο για να γίνει κάτι. Πάντοτε η κάθε χώρα θα πρέπει να ασκεί πίεση στη δική της κυβέρνηση, όπως ας πούμε η Βουλγαρία. Θα ασκεί ε, πίεση ώστε να περνάνε στο Συμβούλιο ε, οι αντίστοιχες γραμμές, ε, π.χ. η έγκριση και κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αλλά και το θέμα της πάταξης της βίας κατά των γυναικών. Τώρα, πάμε στο τρίτο πάνελ που είναι ο δρόμος προς την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Να δούμε λίγο τα μέλη του πάνελ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ. Είναι η αρχή της τελευταίας ε, συζήτησης πάνελ αυτή. Να προσκαλέσω λοιπόν τους επόμενους ομιλητές. Πρώτη η κυρία Λίζα Οβλίρ από το Ιστονικό Κοινοβούλιο, μετά η κυρία Γκουλσούν και Κεχάν από το Συμβούλιο της Ευρώπης και η κυρία Λάουρα Άλμπου από το Ευρωπαϊκό Λόμπι των Γυναικών. Παρακαλώ.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 is she has even mentioned this time she said that. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ξεκινάμε με το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας συζήτησης. Τον λόγο έχει πρώτη η κυρία Λίζα Όβιρ η οποία είναι μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Εστονικού Κοινοβουλίου. Έχετε 7 λεπτά, παρακαλώ. Chair. Κυρία Πρόεδρε, μέλη των Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία και για την πρόσκληση καθώς μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Θα συνεχίσω στα εστονικά, την πανέμορφη μητρική μου γλώσσα. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2011 η Εστονία υπέγραψε το Δεκέμβρη του 2014. Προσφάτως μόλις, στα τέλη Σεπτεμβρίου φέτος, το Εστονικό Κοινοβούλιο κύρωσε τη σύμβαση. Η σύμβαση βασικά έχει ως στόχο να μας δώσει μια Ευρώπη στην οποία δεν έχει θέση βία κατά των γυναικών, σε οποιαδήποτε μορφή της. Το νομικό πλαίσιο λοιπόν πρέπει να προστατεύει τις γυναίκες από τη βία και να ε, εισαγάγει την ισότητα των δύο φύλων. Πολύ συχνά βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτό αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα και όχι πρόβλημα της συγκεκριμένης οικογένειας. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ζήτημα και στην Εστονία. Το 50% του πληθυσμού μας έχουν είτε ακούσει, είτε έχουν δει, είτε έχουν βιώσει άμεσα ενδοοικογενειακή βία. Παρόλο που ο κόσμος καταδικάζει την ενδοοικογενειακή βία, το 10% εξ αυτών θεωρούν ότι κάποιες φορές είναι απαραίτητη. Πολλές φορές ε, βέβαια βλέπουμε και την τάση να κατηγορείται το θύμα. Το 14% των αισθανών θεωρούν ότι εν μέρει φταίνε και τα θύματα για την ενδοοικογενειακή βία. Στο 70% των περιστατικών οι δράστες είναι σύντροφοι ή πρώην σύντροφοι. Στο 80% των περιστατικών οι δράστες είναι άντρες και τα θύματα συνήθως γυναίκες. Πολλές ε, μελέτες έχουν γίνει στην Εστονία μέσα στα πλαίσια της σύμβασης. Σε μια μελέτη που έγινε για την ενδοοικογενειακή βία το 2011 είδαμε πως το 12% των γυναικών στην Εσθονία είχαν βιώσει σεξουαλική βία στο σπίτι τους, σωματική και σεξουαλική βία. Όσον αφορά στη σεξουαλική βία, είχαμε 10.000 γυναίκες και 12.000 για την σωματική βία. Είναι ζωτική σημασία να υπάρχουν χώροι όπου οι γυναίκες μπορούν να καταφύγουν όταν πέσουν θύματα ή πριν πέσουν θύματα για να μπορέσουν να μην έχουν πλέον βία στη ζωή τους. Το 2016 έγινε και μια μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με την οποία η βία αυτή στοιχίζει στην κοινωνία και στο κράτος πολλά, διότι υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, το σύστημα της δικαιοσύνης που εμπλέκονται, αλλά φυσικά τα θύματα, τα ίδια τα θύματα, έχουν σοβαρές επιβλαβείς επιπτώσεις μεταξύ άλλων στη σωματική και ψυχική τους υγεία. Επίσης υπάρχουν μεγάλες απώλειες ε, για τους εργοδότες. Το κόστος της ενδοοικογενειακής βίας στην Εστονία λοιπόν υπολογίζεται στα 116 ευρώ ανά έτος, για να μην να αναφέρουμε και όλες τις ζωές που έχουν καταστραφεί την ίδια στιγμή. Στις αρχές του 2017 η κυβέρνηση κατέθεσε στο Κοινοβούλιο τη Σύμβαση Προσκύρωση. Έγιναν κάποιες ε, αλλαγές νομοθετικές όσον αφορά τον κώδικα για τις εφέσεις ε, αλλά και για την προστασία των θυμάτων. Οι αλλαγές που έχουν να κάνουν με την προστασία θυμάτων περιλαμβάνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στα κέντρα υποστήριξης και ε, ως αποτέλεσμα όλων αυτών υπάρχει καλύτερη πρόσβαση σε αυτά τα κέντρα και καλύτερη χρηματοδότηση αυτών των κέντρων. Επίσης υπήρξε μια σειρά δικημάτων που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον ποινικό κώδικα της Εσθονίας ως αποτέλεσμα της ε, σύμβασης. Για παράδειγμα, η επίμονη παρακολούθηση, η ψευδής, συλλευκή λευκή γάμη, η, ο ακροτηριασμός ε, των γεννητικών οργάνων, των γυναικών, πράγματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι κάτι ε, που έχω ζήσει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων προσωπικά. Μελετώντας τη σύμβαση λοιπόν και το σχέδιο της νομοθεσίας, στην ουσία είχα μία ευκαιρία να αναλύσω την κατάσταση που υπάρχει ε, σε νομοθετικό επίπεδο στην ε, Εστονία. «53% των γυναικών ηλικίας άνω των 65 ετών έχουν βιώσει τουλάχιστον μία φορά τη σεξουαλική παρενόχληση στη ζωή τους». Αυτό περιλαμβάνει βέβαια Ε, ε, διάφορες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης όπως ας πούμε το άγγιγμα χωρίς τη θέληση της γυναίκας. Ε, η σεξουαλική παρενόχληση είναι εκτεταμένη και σε κάποιο βαθμό αποδεκτή στην Εστονία, όμως ξεκάθαρα υπάρχουν επιπτώσεις για το θύμα, την υγεία του και την ιδιωτική του ζωή. Μόνο μία υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Αυτό για μένα σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ρύθμιση σε αυτό το τομέα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομοθεσία, οι γυναίκες στην ουσία δεν είχαν προστασία, γιατί δεν υπήρχε και δεδικασμένο. Η ρύθμιση λοιπόν του ζητήματος αυτού, ε, της σεξουαλικής δηλαδή παρενόχλησης μέσω της νομοθεσίας ε, ήταν ζωτική σημασία. Μετά τις ε, πρώτες αλλαγές στην νομοθεσία είχαμε και τις πρώτες καταγγελίες στην αστυνομία. Η κύρωση στα τέλη της Σεπτεμβρίου είναι απλώς η αρχή. Το Ιστονικό κράτος έχει καταδείξει τη δέσμευσή του να προστατεύει τις γυναίκες, τα θύματα και να αντιμετωπίζει κατάλληλα τους δράστες. Το ζήτημα έχει συζητηθεί ευρέως στην Εστονία. Ξέρω ότι παρά το γεγονός ότι έχει γίνει ένα τεράστιο άλμα προς την ε, ε, ε προς την ε, ευαισθητοποίηση θα έχουμε κάνει και ένα τεράστιο βήμα και προς την σωστή κατεύθυνση για το θέμα αυτό. Τώρα έχει το λόγο ε, η κυρία από το, Ευρωπαϊκό, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η κυρία Γκουλσούν Μπιλγκεχάν, Γενική Εισηγήτρια για τη Βία κατά των Γυναικών. Merci, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι υπάρχουν πιο πολλές γυναίκες και, και λιγότεροι άνδρες στην αίθουσα, αλλά είναι λογικό όταν μιλούμε για ζητήματα ισότητας, ε, γιατί συνήθως σε εμάς αφορά. Είναι τεράστια χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να έχω τη δυνατότητα να ε, συζητήσω μαζί σε αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους η καταπολέμηση των, ε, της ε, βίας που υφίστανται οι γυναίκες το βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το περασμένο Ιούνιο είναι ένα εξαιρετικά θετικό βήμα είναι ένας επιπλέον λίθος στο οικοδόμημα ένα οικοδόμημα που σκοπό έχει να εξαλείψει κάθε είδους βία στην κοινωνία μας Ασχολούμαστε από τον Οκτώβριο, ε, ασχολούμαι από τον Οκτώβριο του 2017 ως Γενική Εισηγήτρια για το θέμα αυτό ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ασχολούμαι επίσης με το θέμα της καταπολέμησης της βίας των γυναικών εδώ και πολλά χρόνια. Ε, έχω ασχοληθεί με μια έκθεση που αφορά την παρενόχληση ε, των γυναικών σε δημόσιους χώρους, όπως επίσης και με τους εξαναγκαστικούς γάμους. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε ακόμη να κάνουμε για την ε, βία κατά των γυναικών. Αν υπάρξουν ε, ειδικέ νομοθεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτό δεν αρκεί, είναι πολύ πιο εκτεταμένο το πρόβλημα και οι νοοτροπίες εξελίσσονται πολύ αργά. Εγώ είμαι βουλευτής της Τουρκίας. Η χώρα μου ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε και επικύρωσε ε, την σύμβαση αυτή, άλλωστε εξού και σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Μερικές φορές είναι εύκολο, εντάξει, όχι εύκολο, αλλά χρειαζόταν πολύ ε, ε είναι πολύ σημαντικό και μετά για την εφαρμογή ε, της σύμβασης αυτής να υπάρχει ε, σθένος. Όπως είπε ο ανθρωπολόγος και επίτιμος καθηγητής ε, Φρονσουά ο οποίος ε, απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα, Μιλάμε για μια φύση η οποία θα ήταν βίαιη η φύση των ανδρών και η οποία είναι κυριαρχική εκφύσεως. Μιλάμε επίσης και για βιαιοπραγίες, για θηριωδίες. Ε, όχι, δεν είναι εκφύσεως το πρόβλημα, είναι μια κουλτούρα αυτή που δημιουργεί αυτή τη βία. Και ε, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το θέμα της κουλτούρας, της σκέψης, ε, της, ε, του, τρόπου σκέψης μας, μπορεί ο αγώνας μας να αλλάξει την κουλτούρα αυτή εμείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, όταν θέλουμε να ε, καταπολεμήσουμε τη βία δεν θέλουμε απλώς να εξυπηρετήσουμε την ιδεολογία ε, των φίλων και να καταστρέψουμε την οικογένεια. Μετά την έναρξη ισχύω σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ο αγώνας άρχισε να έχει ένα επιπλέον όπλο στο πλωστάτιό του, στο πλωστάσιό του δηλαδή τα κράτη-μέλη μπορούν πλέον να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τις σχετικές αλλαγές και να γίνει ένα νομοθετικό μέσο. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αναγνωρίζει τη βιαιότητα κατά των γυναικών ως μορφή διάκρισης και ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέτει το θύμα στο επίκεντρο κάθε μέτρου που πρέπει να ληφθεί. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της πρόληψης, της προστασίας των θυμάτων και της τιμωρίας των θητών ε, πρέπει να συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε ως ε, προς το πόσο επίγον είναι να ε, καταπολεμήσουμε και να προβλέψουμε τη βία κατά των γενικών και πρέπει οι ε, αρχές να υποστηρίξουν τα θύματα μέσω της εφαρμογής της αποτελεσματικής της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δίνει ένα διεθνές πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό οι βουλευτές έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Μέσω του άρθρου 70 η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δίνει ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια πολύ σημαντικό ρόλο, καλώντας τα να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής της. Είναι η πρώτη φορά που ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στην παρακολούθηση αναφέρεται ρητά σε, σε μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που τίθεται. Τι μπορεί, πώς μπορούν τα ε, κοινοβούλια να συμμετέχουν ε, ενεργά στην παρακολούθηση της σύμβασης και να εξασφαλίζουν ότι ε, εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Πρώτον, πρέπει να υπενθυμίσουμε τον πρωταρχικό ρόλο των εθνικών βουλευτών, που είναι η ψήφιση της νομοθεσίας, που έχει ένα άμεσο αντίκτυπο ως προς την ε, εφαρμογή της, ε, της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ε, γιατί πρέπει να είναι σύμφωνη η εθνική νομοθεσία με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριμένη σύμβαση. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρξουν προσαρμογές αν χρειάζεται της εθνικής νομοθεσίας, να υπάρχουν μέτρα προσαρμογής δηλαδή για να συνάδει η ένομη τάξη του κράτους, του συμβαλωμένου κράτους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση σύμβαση. Επίσης, ο προϋπολογισμός είναι κάτι το οποίο ε, εγκρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ένα οικονομικό αντίκτυπο οι περισσότερες ε, διατάξεις της σύμβασης, όπως για παράδειγμα τα καταφύγια για τις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Ε, λόγω λοιπόν του ρόλου τους προς την έγκριση του προπολογισμού του κράτους, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν και πάλι ένα μοχλό ε, πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο προϋπολογισμός τους δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν ότι τα μέσα που διατίθενται για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι επαρκή. Η παρακολούθηση από τους βουλευτές περνά και από τον έλεγχο της δράσης της κυβέρνησης. Και εγώ από την αντιπολίτευση προέρχομαι. Για να γίνει αυτό υπάρχουν πολλά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, εμείς ως βουλευτές, για παράδειγμα ε, παρουσία του αρμοδίου υπουργού κατά τις δημόσιες συζητήσεις, ε, ε, που πρέπει να ενημερώνεται για τα μέτρα της κυβέρνησης ε, ώστε να συμμορφώνεται η χώρα με τις υποχρεώσεις εκ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Συμβούλιο της Ευρώπης είχε ζητήσει τη δημιουργία δομών συγκεκριμένων ειδικών στο πλαίσιο των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπως οι επιτροπές ε, που είναι επιφορτισμένες με ζητήματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι δομές πρέπει να εξασφαλίσουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο, τακτικό έλεγχο, του σεβασμού των διεθνών υποχρεώσεων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμω, πρέπει να τεθούν τα ερωτήματα και πρέπει να υπάρξουν και απαντήσεις. Ένα ακόμα ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ε, το 2014 είχε τονίσει τη σημασία τα εθνικά κοινοβούλια να ζητούν ε, την άποψη εθνικών ιδρυμάτων ε, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό τα κοινοβούλια να έρχονται σε διάλογο και με εξειδικευμένα ιδρύματα αλλά και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία γιατί έτσι θα έχουν ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη στη διάθεσή τους που θα τους δίνει τη δυνατότητα να ε, παρακολουθήσουν αποτελεσματικά την εφαρμογή της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Η επίβλεψη της εκτελεστικής εξουσίας όμως δεν είναι πάντοτε επαρκής. Πρέπει και το Κοινοβούλιο να συμμετέχει απευθείας στις εκθέσεις. Το άρθρο 70 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης εξασφαλίζει στα Εθνικά Κοινοβούλια την πρόσβαση ε, στους μηχανισμούς αξιολόγησης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της εφαρμογής της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν αυτό τον ρόλο στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης ε, από τις κυβερνήσεις. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω Λέγοντα ορισμένα πράγματα για τα ε, δίκτυα των κοινοβουλίων ε, ε, για τα θέματα γυναικών, τα οποία συντονίζω. Σήμερα το πρωί είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για το θέμα αυτό με εμπειρογνώμονε και βουλευτές. Για να ολοκληρώσω, τα έχουμε πει σχεδόν όλα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι χάρη στη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, η βία κατά των γυναικών καταδικάζεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό και διεθνές ε, σε όλες τις πτυχές της. Πρέπει όμως να την εφαρμόσουμε και πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την βία κατά των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, και τώρα η κυρία Λάουρα Άλμπου. Έχετε το λόγο. For Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την πρόσκληση αυτή της στα πλαίσια της Διεθνούς ημέρας κατά της βίας κατά των γυναικών. Θα ξεκινήσω παρουσιάζοντας ε, το European Women's Lobby, η μεγαλύτερη συνομαδοποίηση μη όμικρον ομάδων πιέσεων από όλη την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την ε, Σερβία και την ε, Μακεδονία εγώ προέρχομαι από, το, από την αντίστοιχη Ομοσπονδία Ενώσεων της Ρουμανίας, φορέας ε, που έχει πρωτοστατήσει στην συλλογή δεδομένων και στην ευαισθητοποίηση προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι υψηλή προτεραιότητα η αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε μια διεπίπεδη πραγματικότητα. Φαίνεται ότι καταρχάς τα αιτήματα των ενώσεων γυναικών λαμβάνονται πλέον σοβαρά υπόψη και έχουμε δει και εξελίξεις στις λήψεις αποφάσεις για τις πολιτικές μία από τις ενδείξεις ε, της πρόοδου αυτής είναι και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολη η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με συγχωρείτε το 2017 επελέγει ως έτος για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και είναι και βεβαίως και η, ημερομηνία των υπογραφών της συμβάσεως. Μετά την έγκριση της πλατφόρμας για δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλει ένα ισχυρό, <clears throat> ισχυρό με μήνυμα για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών και την ανάληψη νομοθετικών και άλλων μέτρων. Όμως, και αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο της πραγματικότητας, πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Έχουμε πολλά κενά τα οποία έχουν παρουσιαστεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι οι 35 εμπειρογνώμονές μας του δικτύου της ε, Ένωσης του Λόμπι των Γυναικών βλέπουμε ότι η προστασία που λαμβάνουν οι γυναίκες είναι πάρα πολύ διαφορετική διαφοροποιημένη εντός της Ευρώπης υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ της προστασίας και των δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη. Τα διάφορα ψηφίσματα υπέρ των γυναικών συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου το Σεπτέμβριο πολύ ισχυρού ψηφίσματος με συντριπτική πλειοψηφία φτάνουν συνεχώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ανάλογα με το πού είναι κάτοικος η συγκεκριμένη γυναίκα μπορεί να μην έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν γραμμές ΣΟΣ σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γραμμές εκτάκτου ανάγκης, τηλεφωνικές δηλαδή. Δεν έχουμε επαρκή δεδομένα και δεν ξέρουμε πόσες ακόμα γυναίκες θα πρέπει να δολοφονηθούν ή να βιαστούν προτού η Ευρωπαϊκή Ήπειρος αποφασίσει ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα και μη ανοιχτά. Γι' αυτό προχωρήσαμε στην, στο σχηματισμό μιας συμμαχίας για την προστασία των ενδομένων των ανηλίκων αλλά και άλλων μειονοτήτων, των ηλικιωμένων, των ε, ε ανθρώπων διαφοροποιημένου σεξουαλικού προσανατολισμού. Ε, η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται πλέον άμεσα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι που κατοικεί στην Ευρώπη θα μπορέσει να έχει να της εξασφαλιστεί ότι θα έχει μια ζωή χωρίς βία κρούσματα, χωρίς να υφίσταται δηλαδή βία που θα της υφίσταται απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκα. Υπό τις πρωτοβουλίες επίσης της Εστονικής Προεδρίας συνεχίσαμε την όθηση αυτήν για να εξασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση επικύρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμβασης Κωνσταντινούπολης και προκειμένου να εγκρίνουμε έναν κώδικα δεοντολογίας πανευρωπαϊκά. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό θέμα το οποίο επομένω απαιτεί πανευρωπαϊκή απάντηση. Τώρα έχουμε μια ευκαιρία για να δουλέψουμε συλλογικά ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις πιο σημαντικές διατάξεις της σύμβασης. Την προστασία δηλαδή των θυμάτων και τη δίωξη και τιμωρία των θητών. Επομένως η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να πάει πέραν της συζήτησης προκειμένου να επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και, και, και προκειμένου να αποσαφινιστούν οι μικτές ή άλλες αρμοδιότητες. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσει στους επόμενους μήνες τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με το ευρύτατο δυνατό πεδίο ερμηνείας Ελπίζουμε λοιπόν ότι και οι επεργόμενες προεδρίες της Βουλγαρίας και της Αυστρίας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν ότι αυτό θα γίνει έγκαιρα. Καλούμε ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης εδώ και 20 χρόνια. Τώρα με ικανοποίηση βλέπουμε κάποια θετικά βήματα αλλά περιμένουμε πραγματικές αλλαγές, όχι απλές δηλώσεις. <clears throat> Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωριστεί από Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών ότι υπάρχει μια σειρά κρουσμάτων που ασ... αβίας που ασκούνται από τους άνδρες κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες. Τι άλλο ζητούμε. Μια συνολική στρατηγική, μια συνολική πολιτική παροχής βοήθειας στα θύματα, γιατί χωρίς τη στρατηγική, χωρίς τις πολιτικές δεν θα υπάρχει προϋπολογισμός και κυρίως δεν θα υπάρχει προϋπολογισμός και οικονομική βοήθεια για τις ε, πολιτικές που αφορούν στην ισότητα των φύλων. Ζητούμε λοιπόν να διοριστεί ένας Ευρωπαίος συντονιστής όλων των πολιτικών για την εντόπιση αυτών των κρουσμάτων βίας, ώστε να συντονίσει μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών, υπηρεσιών και εθνικών πολιτικών. Επίσης ζητούμε συστηματική διαβούλευση και συστηματική χρηματοδοτική στήριξη της ενώσεις υπέρ των γυναικών και των κοριτσιών, όπως και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως και σε τοπικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εψήφισε, όπως έλεγα το Σεπτέμβριο, με συντηρητική πλειοψηφία, με ευρύτατη στήριξη διαμέσω διαφόρων πολιτικών ομάδων, για την υιοθέτηση των πολιτικών αυτών, την ε, επικύρωση της συμβάσεως της Κωνσταντινούπολης και την ανάληψη άλλων νομοθετικών μέτρων. Θα ευχαριστούσαμε τις συνεισηγήτριες Μαρία Κοράτσα και την κυρία Μποναφό για την εξαιρετική δουλειά τους. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι μια σαφής αφηρημένη έννοια. Μιλούμε για συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις, τις οποίες έχουμε τονίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια Τη προσπάθειάς μας. Πρέπει οι φωνές των γυναικών να ενισχυθούν ώστε να μην μπορούν πλέον να αγνοούνται. Όπως είχε πει μία φεμινίστρια, δεν υπάρχει καμία γυναίκα που να μην έχει φωνή. Υπάρχουν μόνο εκείνες που επίτηδε τις αγνοούν. και μιλούμε εδώ και για γυναίκες που δεν κατέχουν έγγραφα ταυτότητας, πρόσφυγες, μετανάστες. Πρέπει να είμαστε πλέον θαραλέοι και προκειμένου να αναλάβουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ώστε αυτές οι δηλώσεις να γίνουν πραγματικότητα. Και θα ήθελα επίσης να σας καλέσω να συμμετάσχετε στην ε, διακήρυξή μας ε, για την υπογραφή της συμβάση τη Κωνσταντινούπολη, στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Γερμανικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινή πρωτοβουλία με το Συμβούλιο τη Ευρώπη, Παρακολουθήστε μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωση για αυτό το διάστημα που αφιερώνεται στην καταμολέμηση της βία κατά των γυναικών. Και όπω λέει η κονκάρδα μου, δεν θα περιμένουμε άλλον έναν αιώνα, ήρθε η στιγμή. Και τώρα e, έχουν το λόγο οι συγητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ, πρώτη για πέντε λεπτά, όχι παραπάνω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετική ευκαιρία, μια σημαντική ευκαιρία σήμερα όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα εθνικά κοινοβούλια. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μια ευθύνη για την κύρωση της σύμβασης ε, της ε, Κωνσταντινούπολης. Ε, πραγματικά το Συμβούλιο της Ευρώπης οφείλουμε τη σύμβαση και ευχαριστώ Λάουρα που μας έδωσες την ε, αίσθηση του πόσο επίγον είναι αυτό το θέμα και σε ευχαριστώ που μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα η σύμβαση να εφαρμοστεί στην πραγματική, την καθημερινή μας ζωή. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα ακόμα είναι ε, ευρέως διαδεδομένα και γίνονται ανεκτά στην Ευρώπη. Σήμερα δίνουμε μια φωνή σε εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια που η ζωή τους έχει καταστραφεί από τη βία τους λέμε δυνατά και φωναχτά ότι δεν είναι μόνες τους και ότι νοιαζόμαστε για αυτές. Επίσης σε δημόσιους χώρους, ε, στο σπίτι μας αλλά και στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε ένα νέο ε, παγκόσμιο φαινόμενο όπως ε, και νέα εγκλήματα. Η πορνογραφία ως εκδίκηση, πράγματα δηλαδή που καταστρέφουν ζωές. Αναφέρατε το μητού. Είναι ένα φαινόμενο εκπληκτικό, διότι μας δείχνει πώς είναι η παρονόχληση στον εργασιακό χώρο. Ευρέως διαδεδομένη. Λίγο πολύ όλοι τα ξέραμε αυτά. Όμως έχουμε μείνει άφωνοι από την ευρύτητα του φαινομένου και από το πόσες γυναίκες πριν από 20-30 χρόνια, αλλά ακόμη και σήμερα, υποφέρουν από την κατάχρηση ισχύω και εξουσίας ε, που έχουν οι άντρες στα χέρια τους. Ήρθε η στιγμή λοιπόν οι γυναίκες να υψώσουν τη φωνή τους, να μιλήσουν δυνατά και να καταδικάσουν. Όταν καταδικάσεις ε, δεν υπάρχει δυστυχώς ε, υποστήριξη. Όταν έχεις περάσει από αυτή την ντροπή και την έκθεση γιατί ακόμα πολλές φορές και οι ίδιες οι γυναίκες δεν σε λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Γιατί έτσι είναι το περιβάλλον, αυτά πρέπει να κάνεις, αυτά πρέπει να περάσεις. Ε, σου λένε, αν θέλεις να έχεις μια δουλειά, αυτό είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μιλάει για την ποινικοποίηση μεν, αλλά μιλάει και για την αλλαγή της ονοτροπίας, την πάταξη των στερεοτύπων σε μια κοινωνία η οποία χρειάζεται μια κουλτούρα σεβασμού για τις γυναίκες και τα κορίτσια, η οποία θα εμπλέκει τους άντρες και τα γόρια. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε το βάρος της ευθύνης και της ντροπή να πάει από το θύμα στο θήτη. Να μην έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι, αισθάνονται ένοχες, που τις κάνουν να αισθάνονται ένοχες και ζουν στην ντροπή και την απομόνωση. Στη δεκαετία του 90 στη Σουηδία είχαμε ένα κίνημα κατά το οποίο εκατοντάδες ηθοποιοί σε όλα τα θέατρα της Σουηδίας διάβαζαν φωναχτά ιστορίες γυναικών θυμάτων. Το θέμα και το σύνθημα ήταν ότι δεν θα συγγίσουμε άλλο να σας πω ότι δεν κοιμόηθηκα όλη νύχτα παρόλο που τα ήξερα όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενισχύσουμε τις γυναίκες, να τις κάνουμε να σπάσουν τη σιωπή, να καταδικάσουν, να πάνε στην αστυνομία, στις αρχές, να αισθάνονται εμπιστοσύνη, γιατί αυτό πρέπει να νιώθουν, ότι αν υπάρχει ποινικό αδίκημα θα τιμωρηθεί. Να υπάρχουν ξεκάθαρες κυρώσεις και οι θύτες να καταδικάζονται. Βέβαια, όπως ακούσαμε, τις περισσότερες φορές οι άντρες είναι οι είναι η ζήλια, η ματέωση, το αλκοόλ, επειδή δεν του υποτάσσεσαι, είσαι πολύ ανεξάρτητη, πολύ σύγχρονη, πολύ διαφορετική, πολύ δυνατή. Να αναφέρω και κάτι για τα εγκλήματα τιμής τις δολοφονίες αυτές, τις απεχθείς δολοφονίες, γιατί υπάρχει η συνέργεια των ίδιων των γυναικών, της φατρίας, ε, της φιλής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τα γνωρίζουμε αυτά. Δηλαδή, κανένας λόγος δεν υπάρχει για να δικαιολογήσουμε τη βία, ούτε η θρησκεία, ούτε η κουλτούρα και ο πολιτισμός είναι διαφορετικές ερμηνείες της θρησκείας που μας οδηγούν στην καταπίεση και την βία κατά των γυναικών. Εγώ και η συνάδελφός μου η Κριστίν έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας, έχουμε ενώσει τις πολιτικές ομάδες, αλλά και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να προσχωρήσουμε στη σύμβαση. Γιατί γιατί χρειαζόμαστε μια εργαλειοθήκη που να μην είναι τόσο περιορισμένη. Θέλουμε κοινά εργαλεία, ισχυρά εργαλεία και δυνατότητα εφαρμογής. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι, παρακαλώ, ας κάνουμε όλοι μαζί περισσότερα πράγματα για να κυρώσουμε να πείσουμε τη Γερμανία και άλλες τόσες χώρες που δεν έχουν κυρώσει. Όπως είπατε, έχουμε ένα θέμα με την λανθασμένη κατανόηση του ορισμού του φίλου. Ζητώ από τους συναδέλφους στο Συμβούλιο της Ευρώπης να μας βοηθήσουν γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για τη βία κατά των γυναικών, βία που διαπράττεται μόνο και μόνο επειδή αυτές είναι γυναίκες. Θέλω όλοι μαζί να πούμε ότι θα υπάρχει μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Κοράτσα Μπίλτ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κριστίν Ρεβόντα Λόγμπον για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ τις προσκεκλημένες και όλους τους βουλευτές, ευρωβουλευτές και εθνικούς βουλευτές για να δείξουν πόσο κοινό είναι το ενδιαφέρον μας για να δράσουμε επιτέλους. Επιτέλους λύνεται η γλώσσα μας και μπορούμε να αναλάβουμε μια ευθύνη που είναι τεράστια. Με την Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ είμαστε συνεισηγήτριες για την υπογραφή και την προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πραγματικά επίγον και απαραίτητο τώρα που έγινε υπογραφή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει και η κύρωση ώστε να είναι πλήρως εφαρμόσιμη, ώστε οι τρεις πυλώνε, η πρόληψη, η προστασία και κυρίως η συνέχιση, α, συγγνώμη, δίωξη των ε, ε, εγκληματιών να ε, ισχύουν και οι τρει, Το να υπάρχει δηλαδή υπογραφή χωρίς κύρωση δεν μπορούμε να δράσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης βρισκόμαστε τώρα σε μία περίοδο που είναι πάρα πολύ σημαντική εργασίας, συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, για τους ε, κώδικες δεοντολογίας, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό να ε, δράσουμε από κοινού. Νομίζω ότι είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο πρώτης υπογραφή, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Έχουμε μία πλήρη αρμοδιότητα ε, για τα διάφορα ζητήματα που καλύπτει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ώστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ακόμη και αν δεν έχουν κυρώσει όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την προστασία σε, όλα, σε όλες τις γυναίκες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Ευρωβουλευτές να ενημερώνονται για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και να μπορέσουμε να, συνο... να, μπορέσουμε να τους, να τους ε, βοηθήσουμε στην προσπάθειά τους. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ ε, την Εστονία που πολύ προσφάτως ε, κύρωσε την σύμβαση. Η Εστονική Προεδρία ε, πίεσε πάρα πολύ. Ελπίζουμε η Βουλγαρική ε, Προεδρία να κάνει το ίδιο για να μπορέσουμε να σταματήσουμε μια κατάσταση που είναι απαράδεκτη και αδύνατο να συνεχιστεί. Ο 11 είναι τα κράτη-μέλη που ακόμη δεν έχουν κυρώσει, 11 στα 28 είναι πολλά τα κράτη αυτά, κάτι πρέπει να γίνει. Θα θέλαμε λοιπόν να απευθυνθούμε στα κράτη τα οποία έχουν αρχίσει να ε, αναλαμβάνουν μέτρα αρκετά κατά των γυναικών, όπως στην Πολωνία για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια ψήφισε ένα, ε, ε, υπερψήφισε ένα ψήφισμα για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία, μια έκθεση εξαιρετικά ανησυχητική, στην οποία αναφέραμε ότι τα δικαιώματα των γενικών είναι τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να την χάνουν τη ίδια προστασία στην Πολωνία, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα, και είναι σημαντικό να το επισημαίνουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη όλα να κυρώσουν αυτή τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής, ώστε να υπάρχει ένας κώδικα συμπεριφοράς ε, πλήρης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία νομοθετική πράξη επί της οποίας θα εργαστούμε για να υπάρξει μία ε, γενική οδηγία ε, προστασίας των ε, γυναικών ε, κατά της καταπολέμησης που υφίστανται. Ευχαριστούμε την κυρία Μπονφούα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ, έχετε δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τέλος πλέον της ημέρας ε, της συνειδρίασης, Απλώς θα σας δώσω μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τα όσα συμβαίνουν ε, στην προετοιμασία του κώδικα δεοντολογίας ε, για τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Είχαμε καταρχάς δύο ημέρες συζήτηση στο κολόκουιουμ των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών το θέμα ήταν μεταξύ των πρώτων που χειριστήκαμε. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το επίπεδο φιλοδοξία της Κομισιόν είναι το υψηλότερο που είχαμε ποτέ. Και το επιβεβαίωσε και η Επιτρόπος. Και πραγματικά ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι αυτό, αυτή, αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας θα πρέπει να μετατραπεί σε επικύρωση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα, μια πρόταση κειμένου από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κώδικα διοντολογίας. Το εξετάζει αυτή τη στιγμή η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου υπό την Εστονική Προεδρία. και μας δεσμεύει η υπογραφή της απόφασης όπου δυστυχώς το πεδίο εφαρμογής η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε περιοριστεί από τα κράτη-μέλη μόνο σχετικά με την μεταρρύθμιση των σχετικών διατάξεων για το άσυλο και τα δικαιώματα των θυμάτων. Αυτή η μεικτή αρμοδιότητα, αυτή η περιορισμένη αρμοδιότητα δεν έχει αλλάξει, είναι το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε. Προσπαθούμε όμως η πρακτική υλοποίηση να είναι όσο το τον ευρύτερη, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ομιλεί με ενιαία φωνή δίνοντας κατευθύνσεις και συστάσεις για τις μελέτες του Γκράβιο και άλλων ενώσεων. Η δουλειά αυτή συνεχίζεται στην ε, ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Έχουν λάβει χώρα κάποια δεν μπορώ να σας πω ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκονται τώρα, αλλά προσπαθούμε αυτό να αναπτυχθεί ως πρακτικός οδηγός για τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν, προκειμένου να υλοποιηθεί με το πιο εύκολο δυνατό τρόπο. Χρησιμοποιήσαμε ως πρότυπο τον κώδικα διοντολογίας για τους ανθρώπους με αναπηρίες και τη σχετική σύμβαση ελπίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επικύρωση ελπίζω στους ε, επόμενους λίγους μήνες υπό την Βουλγαρική Προεδρία αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πολλά περισσότερα. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι αυτό δεν πρόκειται να πεπεκτείνει το πεδίο αρμοδιότητας της υπογραφής Απλώς προσπαθούμε η εστίασή μας να είναι όσο πιο πρακτική γίνεται για να πάμε στα της υλοποίησης. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση αυτή, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έξι, έξι ομιλητές έχουμε στον κατάλογο. Όλοι θα έχουν δυνατότητα να παρέμβουν, αλλά δεν μας απομένουν παρά εννέα λεπτά τουλάχιστον Ω προ τη διερμηνία. Οι διερμηνείς θα πρέπει να σταματήσουν στις 6.30. Και αν μας παραχωρήσουν και ένα έξτρα πεντάλεπτο, λέει ο Πρόεδρος, θα είναι ιδιαίτερα ευγενική. Εάν λοιπόν δεν τηρήσετε αυστηρά χρονικά περιθώρια θα σας διακόπτω. Παρακαλώ εκπρόσωπος του Βελγικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη και ίσως να μην μου χρειαστούν καν δύο λεπτά. Να σας πω λοιπόν για την κατάσταση στο Βέλγιο. Εδώ και πολλά χρόνια εμείς έχουμε δεσμευτεί να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και βίας μεταξύ των φίλων. Από το 2001 έχουμε εστιαστεί στην καταπολέμηση των κρουσμάτων αυτών ως ε, μέρος ενός, ενός σχεδίου, σχεδίου δράσεως του οποίου ηγείται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μαζί με τις ε, περιφερειακές αρχές και τοπικές αρχές και συντονίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Ισότιμων Ευκαιριών. Είχαμε διάφορες φάσεις υλοποίησης μέχρι το 3, μετά μέχρι το 7, μέχρι το 9 και μετά από το 10 στο 14 του σχεδίου αυτού δράσεως. Η μεθοδολογία βασίζεται στην ε, αθρηστική βελτίωση των μέσων ε, νομοθετικών και άλλων που έχουμε στη θέση μας για να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά βίας. Παρά τις προσπάθειές μας, το πρόβλημα της βίας ε, κατά των γυναικών είναι ακόμα πολύ σημαντικό για εμάς και γι' αυτό εκινήσαμε ένα πέμπτο πλέον εθνικό σχέδιο δράση το οποίο από το Κοινοβούλιο όπου προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα είδη βίας μεταξύ των φίλων να τα καταπολεμήσουμε και με ιδιαίτερη εστίαση και έμφαση στη σεξουαλική βία. Το σχέδιο δράσης αυτό ευθυγραμμίζεται απολύτως με τη συνθήκη της Λισαβόνας εις ό,τι αφορά στην καταπολέμηση ακριβώς των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής ε, βίας. και εστιαζόμαστε σε όλες τις μορφές βίας όπως σας έλεγα, βία μεταξύ ε, συντρόφων, ε, υπογραφόντων συμφώνων συμβίωσης, ε, σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης. Και το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακολουθήσει μια συνοπτική, μια πλήρη προσέγγιση για το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν ενσωματώσει κάποιες πολιτικές ε, και μέτρα για την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών βίας με ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση και συλλογή δομένων, σχετικά με τα κρούσματα αυτά, την υποστήριξη των θυμάτων, την αποτροπή, την πρόληψη μάλλον των φαινομένων αυτών. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος θα επαναλάβω το, την έκκλησή μου να μην ξεπεράσουμε τα δύο λεπτά. Μιλήσατε πάνω από τρία. Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να είμαστε αυστηροί. Ε, Κύριο Σιμούλη από τη Λιθουανία, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που υπάρχει αυτή η ε, συνάντηση εδώ η οποία στην ουσία ε, ακολουθεί μια άλλη αντίστοιχη συνάντηση στη Λιθουανία ε, κατά την οποία ελέγξαμε τις επιπτώσεις. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας απευθύνθηκε στην Προεδρία και στις στην κυβέρνηση σχετικά με την κύρωση. Η κυβέρνηση έλαβε ήδη την απόφαση και αυτή τη στιγμή το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της Προεδρίας. Δυστυχώς πρέπει να γίνει και αλλαγή της νομοθεσίας ε, και να ληφθούν αποφάσεις μόνο κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ε, ε, απεχθές. Είχαμε κάποιες εμβληματικές περιπτώσεις βίας και έτσι έγιναν κάποια πράγματα. Εκ των προτέρων είναι ξεκάθαρο ποιος κάνει τι. Υπάρχει δηλαδή ένα αναλυτικό ε, δικονομικό και δικαστικό πλαίσιο, όμως δεν υπάρχει χρηματοδότηση, όπως είπαν οι και οι συνάδελφοι. Έχουμε δύο επιλογές. Η Προεδρία ε, ενδεχομένως να απευθυνθεί στο Συνταγματικό Συμβούλιο ή ε, και να γίνει κύρωση της σύμβασης με κάποιες ε, παρεκκλήσεις, κάποιες αποκλήσεις. Ποιες είναι αυτές όμως, γιατί υπάρχουν και άτομα στο κοινοβούλιο μας ε, που στην ουσία επικρίνουν αυτή τη σύμβαση. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει, ε, έχει ο κύριος Γιάν Ρενόφσκι από το Πολενικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση ήταν τελείως ασύμμετρη. Έγινε μια συζήτηση στην Πολωνία και συνεχίζει σχετικά με δύσκολα θέματα ως αποτέλεσμα αυτής της σύμβασης. Ακριβώς επειδή υπάρχει φόβος ότι αυτή η σύμβαση μαζί με πολλά άλλα ε, περιλαμβάνει όχι μόνο στοιχεία θετικά αλλά περιλαμβάνει και απειλές ε, που οδηγούν στην ε, διάλυση της οικογένειας. Οι πολωνικές οικογένειες προστατεύονται από το Σύνταγμα. Τι είναι η πολωνική οικογένεια, είναι ε, η ένωση συζυγική με τα συζυγικά δεσμά ενός άντρα με μία γυναίκα. Αυτό που δεν έχουμε στην Πολωνία είναι ε, η δυτικού τύπου οικογένεια με τα σύμφωνα. Ε, μια σύμβαση στην οποία ε, κυριαρχεί ο άντρας. Εδώ συζητούμε για τη βία. Όμως, η Λίσσα Βίερ έθεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων αναφερόμενη στην οικονομική βία. Αυτό το κομμάτι της σύμβασης το χαιρετίζω. Υπάρχει όντως πρόβλημα οικονομικής βίας σε πολλές χώρες του κόσμου. Φαίνεται με πολλούς ε, τρόπους. Στην Πολωνία 400 εκατομμύρια ευρώ καταβάλλονται σε ανθρώπους ε, που κρύβουν σε διάφορες ευρωπαϊκές ε, χώρες ε, τα χρήματά τους για να διαφύγουν των υποχρεώσεών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε εναρμόνιση και συντονισμό για να αντιμετωπίσουμε αυτή την οικονομική βία και γι' αυτό θεωρώ ότι θα ήταν καλό να κάνουμε εδώ το δεύτερο βήμα της σύμβασης. Ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο η Κλοντέκα Μπούτιτζετ από το Κοινοβούλιο της Μάλτας. Το μέγιστο δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. η ενδοοικογενειακή βία και έμφυλη βία στη Μάλτα αντιμετωπίζεται με ένα νόμο που πέρασε το Μάρτι του 2016. Τον Ιούλιο του 2014 κυρώθηκε η Σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Αυτή τη στιγμή το Μαλτέζικο Κοινοβούλιο συζητά και μια άλλη νομοθεσία για το ίδιο θέμα που θα ενσωματώσει τον νόμο του 2016, θα ενισχύσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, και θα θέσει νέες υποχρεώσεις. Θα υπάρξουν πιο σοβαρές επίσης τιμωρίες για τους θύτες, τους δράστες. Σήμερα μιλήσαμε πολύ για την πολιτική θέληση να ε, μεταφραστούν οι λέξεις ε, σε πράξεις. Πριν από κάποια χρόνια μια γυναίκα σκοτώθηκε, μια γυναίκα γενναία η οποία μίλησε φωναχτά και έριξε φως σε αυτά που ε, ήταν κρυμμένα. Η Ρομπέρτα Μέτσολα ήταν, ε, είχε δεχθεί απειλές και το άτομο που την απειλούσε είχε πάει στο δικαστήριο. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες οι οποίες πάσχουν και υποφέρουν λόγω της σιωπής. Να είναι σίγουρος ότι κάποια μέρα θα έχουν και αυτές δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταία. Ομιλήτρια Άγγελα Γκουέρα από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε κατά την, κατά την καταπολέμηση της βίας ε, μεταξύ των φίλων ε, η Πορτογαλία έχει αναγνωριστεί για τις καλές της πρακτικές. Έχουν υπάρξει εθνικά σχέδια δράσης οποίες ε, τα οποία συνεχίστηκαν ε, από τη μία κυβέρνηση στην άλλη. Έχει αναγνωριστεί ανάγκη επένδυσης ε, στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών μέσω μέτρων προστασίας τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πέμπτο σχέδιο δράσης εθνικό για την καταπολέμηση της βίας της ενδοοικογενειακής. Ξεκινήσε το 2015 και θα εκπνεύσει το Δεκέμβριο του τρέχοντος. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις υποχρεώσεις της Πορτογαλίας στο πλαίσιο πολλών διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων. Και επικεντρώνεται ειδικότερα στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν ε, αναφέρεται μόνο στην ενδοικογενειακή αλλά και σε άλλες μορφές βίας κατά των γυναικών όπως ε, ο ακροτηριασμός γενετικών οργάνων ε, γνωρίζετε όπως υπόθηκε και προηγουμένως από συνάδελφό μου ήταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα μου που ε, ομοφόνος κύρωσε την Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, ε, θέλει να επιτύχει καλύτερη προστασία των γυναικών και τιμωρία των δραστών και καλύτερη κατάρτιση των επαγγελματιών, ε, όπως για παράδειγμα δικαστών, λειτουργών κλπ. Όσον αφορά τώρα την νομοθεσία, έχουν γίνει αλλαγές στον ποινικό κώδικα τον Αύγουστο του 2016 Σύμφωνα με την ε, ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ε, ο εξαναγκαστικός γάμος, η επίμονη παρακολούθηση αναγνωρίστηκαν ως νέα δικήματα, όπως και η σεξουαλική παρενόχληση. Όλα αυτά τώρα έχουν συμπεριληφθεί στην πορτογαλική νομοθεσία, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για την αλλαγή των νοοτροπιών στις ε, διάφορες χώρες. Και βάσει όσων ακούσαμε σήμερα, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη ως προς τη συνεργασία και το συντονισμό. Και αυτό φυσικά είναι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς μας που μας παραχώρησαν πέντε επιπλέον λεπτά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ο τον άλλον. Τελευταία ομιλήτρια για σήμερα. Φαμπρίτσια Τζουλιάνη από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι ήδη περιέγραψαν πόσο σημαντική ήταν η επικύρωση της συμβάσεως στη χώρα μας και πόσο σημαντικό είναι να μετατράψουμε, να μετατρέψουμε τις δεσμευτικές αρχές και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την, ε, τον συσχετισμό μεταξύ της αντιμετώπισης της ανισότητος και των ε, κρουσμάτων που αντιμετωπίζει και διέπει η Σύμβαση θέματα που δεν σχετίζονται μόνο με τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα οποία συμπληρώνουν, ολοκληρώνουν την διαδρομή ελευθερίας που έχουν ακολουθήσει οι γυναίκες στις κοινωνίες μας. Ήθελα απλώς να θυμίσω ότι υπάρχει κάτι απέναντί μας ένα φαινόμενο, ένα κρούσμα όχι μόνο υπόλοιμα της ε, πατριαρχικής ε, κοινωνίας, του συστήματος του πατριαρχικού. Δεν είναι πλέον δηλαδή μια νέα κατάκτηση. Αυτό το έχουμε ήδη κατακτήσει, αλλά πρέπει να προφυλάξουμε τα δικαιώματα που έχουμε κατακτήσει. Πρέπει να τα προασπιστούμε. Δεν είναι κάτι που πλήττει λοιπόν απλώς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πλήττει την συνείδηση, τη δημοκρατική συνείδηση των χωρών της Ευρώπης. Επαναλαμβάνω λοιπόν και εγώ την πρόταση οδηγίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ομαδοποιήσουμε τις διατάξεις αυτές, για να εξωθήσουμε τα κράτη-μόλι να προχωρήσουν προς τα εμπρός και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει την πίασή του ώστε να έχουμε την επικύρωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω ε, τους ομιλητές, τις ομιλήτριες του τρίτου μας πάνελ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Εστονική ε, Προεδρία και την Εστονία που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της κύρωσε τη σύμβαση της ε, Προεδρίας. Ελπίζουμε οι Βουλγαρική και η Αυστριακή να κάνουν το ίδιο. Ευχαριστώ τις δύο συνεισηγήτριες, την κυρία Μπονφουά και την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε που εκφράσατε την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους που των 15 ε, κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής, ε, ε, των, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Νορβηγικού Κοινοβουλίου που τοποθετήθηκαν σε σχέση με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία κηρύξω το πέρα τη ε, συνεδρίαση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στο πλαίσιο άλλων, άλλων διακοινοβουλευτικών ε, ε, συνεδριάσεων να μπορέσουμε να ξαναειδωθούμε. Ευχαριστώ και του διερμηνεί. Σα ευχαριστώ πολύ όλου και ελπίζω να σα ξαναδώ πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη τη Επιτροπή Γυναικών ότι η επόμενη συνεδρίασή μα θα λάβει χώρα στι 4 Δεκεμβρίου στι 3 η ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.